Καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας την απόψινή. Bueno, Ελπίζω να είχατε καλές, μια καλή περίοδο. Και περνάμε στην ημερήσια διάταξη. Σημείο 1 στην ημερήσια διάταξη. Έγκριση του σχεδίου ημερήσια διάταξη. Απλά να σας πω ότι να σας ανακοινώσω ότι σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης διαγράφεται επειδή ο υπουργό ε, Αλληλείας της Νορβηγίας έχει ασθενήσει και δεν μπορεί να έρθει στη συνεδρίαση που είχαμε προβλέψει μαζί της αύριο δηλαδή. Διαγράφεται λοιπόν το 13, διαγράφεται, ακυρώνεται. Και τελευταίο και ζητήσατε τον λόγο. Θέλω να σας πω ότι σε αυτή τη συνεδρίαση θα έχουμε και άμεση διάδοση στο web, στο διαδίκτυο και θα έπρεπε να μιλάτε στο μικρόφωνο το αριστερό σας που έχετε στο αριστερό σας χέρι γιατί διαφορετικά θα υπάρξουν προβλήματα με την ε, τηλεοληψία. Να μιλάτε λοιπόν θα αρχίσω εγώ ίδια να το κάνω, εντάξει, δεν το έκανα, ωραία θα το κάνω. Να το κάνετε κι εσείς, γιατί διαφορετικά η κάμερα δεν θα μπορεί να σας πάρει. Ζήτησε τον λόγο η κυρία Λεβδάν, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. ναι, σας περιμένω. Ja, fru ε. Πρόεδρε, πριν από ένα δεκαπενθήμερο, στην Επιτροπή Ανάπτυξης μας παρουσίασαν ε, μία νομική γνωμοδότηση για τη συμφωνία με το Μαρόκο και τις επιπτώσεις της. Να το δούμε υπό τα διάφορα. Σήμερα. Πώς μπορεί να γίνει. Εντάξει, στην... Ε, υπό τα διάφορα θα το δούμε αυτό, κύριε. Ευχαριστώ. Και έτσι μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 2 της ημερησίας διάταξης, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων 1ης και 2ης Σεπτεμβρίου. Αν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης σήμερα, μεταξύ σήμερα και αύριο, δεν θα υπάρξουν ενστάσεις, θα εγκριθούν. Τρία ανακοινώσει τη Προέδρου. Δεν έχω τίποτα συγκεκριμένο. Υπάρχουν κάποια σημεία, αλλά θα τα εξετάσουμε με τα εξειδικευμένα σημεία της ημερησίας διάταξης. Περνάμε στο 4 λοιπόν αμέσω που είναι το σχέδιο ανάκαμψη, ανάκαμψης, ανασύστασης ε, του Χάλιμπατ ε, στον βορειοδυτικό Ατλαντικό. Απλά, όπως είχα πει και σε προηγούμενη συνεδρίαση, είναι η εφαρμογή, η υλοποίηση της, ε, των κοινοτικών διατάξεων, συστάσεων δηλαδή, που αποφασίστηκαν στη Σολομέλεια της ΝΑΦΟ. Από το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έθεσε ενισχύει μέσω των κανονισμών τάξη και ποσοστώσεων. Είχαμε πει ότι αυτό δεν είναι το πιο σωστό και στις αιτιολογικές σκέψεις ασκώ κάποιες επικρίσεις για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε αυτές τις διαδικασίες να τις μεταθέσει ακολουθώντας τακτικές διαδικασίες και όχι με ανώμαλες διαδικασίες ή ασυνήθιστες διαδικασίες. Αυτή είναι η επίκριση που είχαμε ασκήσει. Αναγνώρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόβλημα και λόγω έλλειψης χρόνου και στελεχών όπως είχε πει, αλλά πρέπει να ακολουθούν οι τακτικές διαδικασίες όπως είπαμε εμείς. Από την άλλη πλευρά είδαμε αν ήταν ε, ευθυγραμμισμένη με τις συστάσεις ε, της ΝΑΦΟ αυτή η πρόταση, είναι εντάξει γιατί διαφορετικά θα υπήρχαν προβλήματα, γι' αυτό λοιπόν δεν κατέθεσα καμιά τροπολογία και συνιστώ να εγκρίνετε την πρόταση της Επιτροπής εσείς. Αν δεν υπάρχει λοιπόν κανένα αίτημα να παρέμβει κάποιος, θα περνούσαμε στην ψηφοφορία αμέσως αυτής της έκθεσης. Λοιπόν, εντάξει, πρώτα απ' όλα λοιπόν ψηφίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εντάξει. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Και ψηφίζουμε τώρα το σχέδιο ψηφίσματος νομοθετικού περιεχομένου. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται ομόφωνα στην επόμενη ολομέλεια θα περάσει του Νοεμβρίου 2. Νοεμβρίου 2, όχι στην πρώτη ολομέλεια, αλλά στην Νοεμβρίου 2. Και περνάμε στο πέμπτο σημείο τη ημερησίας διάταξη, που είναι η πληροφορία τη Ευρω... Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, σε σχέση με την 21η τακτική συνεδρίαση τη Διεθνού Επιτροπής για τη διατήρηση των τονοειδών του Ατλαντικού. Στι 15 Νοεμβρίου τον επόμενο μήνα θα διεξαχθεί η συνεδρίαση αυτή ε, 8 ε, 15 Νοεμβρίου στην Ρεσίφη της Βραζιλίας. Έχετε εγκρίνει τον διορισμό και του κυρίου Ρωμέβα αλλά και εμένα της ίδιας για να παρακολουθήσουμε ως παρατηρητές αυτή τη συνεδρίαση στη Ρεσίφη. Ξέρετε ότι το κυριότερο θέμα το οποίο θα εξεταστεί εκεί, πολλά θέματα θα εξεταστούν και ως κύρια θέματα ιδιαίτερα για τα μεταναστευτικά είδη από, σε σχέση με τον Ατλαντικό και την Μεσόγειο. Αλλά το αστέριο θέμα είναι το θέμα του κοκκινόπτερου τόνου, ερυθρόπτερου τόνου. Έτσι λοιπόν κατά κάποιο τρόπο βλέποντας ποια είναι τα βήματα τα οποία έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από μια πρόταση που έκανε το Μονακό να συμπεριληφθεί στο πρώτο παράρτημα ο ερυθρόπτερος τόνος και υστερότερα τις θέσεις που έλαβαν τα κράτη-μέλη Δεδομένων όλων αυτών, εγώ θα ήθελα επίσης να σας πω ότι σε σχέση με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε είναι μια έκθεση αποτίμησης, αξιολόγησης που έγινε μια συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής που συνήλθε στις 21 και 23 Οκτωβρίου στη Μαδρίτη και συνέταξα μια έκθεση αποτίμησης και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας πληροφορήσει σχετικά και πιο εξειδικευμένα σε βάθος. Επίσης να σας πω και θέλω να το πω δημόσια αυτό, ένα παράπονο που έχω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως πρόεδρος αυτής της Επιτροπής Αλίας και κάνοντας χρήση των αρμοδιοτήτων μου και εξουσιών μου, ζητήθηκε γραπτός ε, στις 14 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους στράφηκα στον κύριο Φωτιάδη που είναι ο Γενικός ε, Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης ε, Μαρίν ζητώντας να μας αποστείλει δύο Την έκθεση αποτίμησης που συντάσσει κάθε έτος η υπηρεσία ελέγχου του Βίγκο και μία έκθεση αποτίμησης. Μία απάντηση πήρα μόνο για τη δεύτερη της έκθεσης, για την έκθεση αποτίμησης της ε, Γενικής Διεύθυνσης ΜΑΡΕ. Αλλά όσον αφορά την έκθεση για τον έλεγχο της υπηρεσίας του Βίγκο που υπάρχει, δεν μου απεστάλλει. Και γι' αυτό θεωρώ ότι, μια και είχα επιμείνει εκ νέου μέσω της γραμματείας να μας αποσταλεί αυτή η έκθεση, Πρέπει να πιέσουμε και να εμείνουμε και θέλω εκπρόσωπο τη Επιτροπής Ξέρω ότι δεν είσαστε εσεί ε, υπεύθυνοι, αλλά είσαστε υφιστάμενοι. Εγώ απευθύνθηκα στον κύριο Φωτιάδη να διαβιβάσετε το παραπονό μου διότι αυτή η έκθεση δεν μας έχει αποσταλεί και αποκρύπτεται. Δεν ξέρω ποια είναι τα προβλήματα. Εγώ συνήθα με τον κύριο Φωτιάδη και είπε ότι θα υπήρχε διαφάνεια με την Επιτροπή μας. Υπάρχει αυτή η έκθεση από την Υπηρεσία Αξιολόγησης και δεν κατανοώ τους λόγους. Αν υπήρχε κάποιος πολύ σοβαρός λόγος και πολύ ευαίσθητος θα μπορούσαν τουλάχιστον να είχαν έρθει σε επαφή με μένα ως πρόεδρο και εγώ θα μπορούσα να αξιολογήσω αν πράγματι για ποιον λόγο δεν διαδόθηκε, δεν ε, μας εστάλει ή όχι. Αλλά να μην υπάρχει μία απάντηση ή μία τελής απάντηση, θέλω να παραπονεθώ και φυσικά αυτό θα το εκλάβω ως μία έλλειψη διαφάνειας για την Επιτροπή μας. Αν δεν πάρω μέσα σε προθεσμία 48 ωρών αυτήν την έκθεση, θα υιοθετήσουμε τα αναγκαία μέτρα και θα απευθυνθώ στον Επίτροπο Μπόργκ για την Αλία με μία, ένα πολύ σοβαρό παράπονο θέλω να εμείνω και να επιμείνω. Δημόσια εδώ το λέω αυτό. Διότι μέσω του ατόμου με το οποίο ήρθα σε επαφή δεν μου δόθηκε η πληροφορία αυτή και θέλω να καταχωρηθεί αυτό το παράπονο. Στη συνέχεια λοιπόν θα, θα δώσω τον λόγο τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο κύριος Βρυμού είναι παρόν παρακαλώ ή όχι. Ποιο είναι εδώ από τη Ευρωπαϊκή επιτροπή που μπορεί να μιλήσει για τον ερυθρόπτερο τόνο, αν κάποιο μπορεί να μιλήσει για αυτό το θέμα. Υπάρχει κάποιο που μπορεί να μιλήσει για τον ερυθρόπτερο τόνο. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ. Δεν ξέρω ποιο είναι, αλλά εσεί έχετε τον... Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι εδώ ο κύριο Γκριμό, η κυρία Ντουάρτε έχει το λόγο ο τόνος ε, και η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Τονοειδών του Ατλαντικού γενικότερα. Η ετήσια συνάντηση αρχίζει ε, την ε, Κυριακή και θα προηγηθεί μια συνάντηση της θερμοστική Επιτροπής της ΕΚΑΤ και όπως όλοι το γνωρίζουν θα είναι πολύ ε, επιβαρημένη η φετινή χρονιά για την ΙΚΑΤ ε, με πολλά αποθέματα για τα οποία θα πρέπει η ΙΚΑΤ να υιοθετήσει ετήσια προγράμματα διαχείρισης, ιδιαίτερα ε, για το απόθεμα του Ξηφία του Βορρά, του Ξηφία του Νότου, και για τον ε, ε, υπέρβαρο τόνο. Ε, για τον τόνο δεν θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε κάποιο σχέδιο φέτος. Έχει υιοθετηθεί ένα νέο σχέδιο από πέρυσι και σιγά σιγά συνηθίζεται αυτό στην ΙΚΑΤ, δηλαδή ο τόνος να καλύπτει τις συζητήσεις και για τη φετινή χρονιά. Θα πρέπει να προσέξουμε λοιπόν πάρα πολύ όσον αφορά το απόθεμα του τόνου και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πολλά άλλα αποθέματα πολύ σημαντικά για τα οποία θα πρέπει να υιοθετήσουμε φέτος ένα σχέδιο διαχείρισης. Η θέση της Επιτροπής που ήδη συζητήθηκε με τα κράτη-μέλη για όλα τα αποθέματα θα βασιστεί κυρίως στη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής. Όσον αφορά λοιπόν τον τόνο, Θέλουμε να ακολουθήσουμε τη γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής που και πάλι δίνει μια σύσταση για μείωση του ΤΑΚ, των συνολικών αλλιευόμενων ποσοτήτων και θα ακολουθήσουμε την γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής. Για τα άλλα στοιχεία του προγράμματος, στο στάδιο αυτό, μπορώ να σας πω ότι ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να ανοίξουμε άλλα στοιχεία. Ένα σημείο κλειδί για μας που πρέπει να το συζητήσουμε για τον τόνο φέτος και πιστεύουμε, επαναλαμβάνω, ότι είναι το σημείο κλειδί για τη διαχείριση και για την αηφορία αυτού του αποθέματος είναι οι δυνατότητες αλίας. Η Επιστημονική Επιτροπή τα τελευταία χρόνια εκφράζει τις ανησυχίες της για την υπερβολική αλλιευτική δυνατότητα που υπάρχει, κυρίως στη Μεσόγειο, για το απόθεμα του τόνου. Και φέτος τα συμβαλόμενα μέρη της ΙΚΑΤ που αλλιεύουν ε, το ανατολικό απόθεμα του τόνου θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΚΑΤ σχέδια διαχείρισης ή μείωσης της αλληλευτικής δυνατότητας. Αυτό κατά μας είναι ένα σημείο κλειδί και θα πρέπει να επιληθεί αυτό το θέμα. Διαφορετικά θα είναι πολύ δύσκολο, για την, ε, θα είναι πολύ δύσκολο να παραμείνει αξιόπιστη η ΕΚΑΤ, όσο δηλαδή υπάρχει υπερβάλλον δυναμικό αλίας. Πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος παράνομης αλίας, αν υπάρχει μεγάλη αλληλευτική δυνατότητα. Ήδη η Επιτροπή έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια για τις αλληλευτικές δυνατότητες και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενότητας που ε, ενδιαφέρονται άμεσα ήδη έχουν κάνει σχέδια σχέδια μείωσης ε, της αλληλευτικής δυνατότητας και τα έχουμε ήδη υποβάλει στην ΙΚΑΤ και ελπίζουμε ότι η ΙΚΑΤ θα ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα της αλληλευτικής δυνατότητας, του στόλου που αλλιεύει τον τόνο για όλα τα συμβαλόμενα μέρη και όχι μόνο για την ευρωπαϊκή κοινότητα. Θέλουμε να παραμείνουμε αυστηρά σε αυτά. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό που ήδη ξεκίνησε φέτος, δηλαδή να εξετάσουμε λεπτομερώς την εφαρμογή της στήρησης των υποχρεώσεων σχετικά με τον τόνο από την Επιτροπή Εφαρμογής. Και αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε το Μάρτιο. Κάναμε μια ειδική συνάντηση της Επιτροπής Εφαρμογής ακριβώς για τον τόνο πολλά προβλήματα εφαρμογής και τήρησης των διατάξεων αναφέρθηκαν και τα συμβαλόμενα μέρη είχαν στη συνέχεια μια προθεσμία για να επιλύσουν τα προβλήματα αυτά. Θα πρέπει να συζητηθεί εκ νέου τώρα στην ΕΚΑΤ. Ελπίζουμε ότι έχουν καταβληθεί προσπάθειες από όλα τα συμβαλόμενα μέρη και ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε σοβαρά αυτή την προσπάθεια και στην επόμενη ετήσια συνάντηση. Λοιπόν, συνοψίζοντας όσον αφορά τον τόνο, τα βασικά σημεία της θέσης μας είναι το ΤΑΚ, το μέγιστο επιτρεπόμενο αλίευμα, σε συνάρτηση με την γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής, η ελευτική δυνατότητα και να καταβληθούν οι απαραίτητες προσπάθειες για να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες που εξέφρασε η Επιστημονική Επιτροπή, και να δοθεί συνέχεια στο σχέδιο ανάκτησης ε, που υιοθετήθηκε πέρυσι, καθώς επίσης και τήρηση όλων των υποχρεώσεων για υποβολή δεδομένων, ε, τήρηση περιόδων αλίας κλπ. Αυτά είναι τα τρία σημεία κλειδιά για μας για αυτή τη συνάντηση της ΙΚΑΤ για τον τόνο. Για τα άλλα είδη, ε, θα σας μιλήσω πολύ σύντομα για τα δύο αποθέματα ξηφία. Η Επιστημονική Επιτροπή επίσης συνέστησε μείωση του ΤΑΚ. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα λοιπόν θα υποστηρίξει τις προτάσεις που θα ακολουθούν την επιστημονική γνωμοδότηση για τη μείωση του ΤΑΚ Και για το Ζεγμονό επίσης η σύσταση είναι μείωση του ΤΑΚ και ένταση της εντατικοποίησης της έρευνας για αυτό το απόθεμα. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τι απόψει τη Επιστημονικής Επιτροπής. Θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε το ΤΑΚ στο επίπεδο που προτείνει η Επιστημονική Επιτροπή. Και επίσης ε, για τον ε, υπέρβαρο τόνο Επίσης, θα ακολουθήσουμε τη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής. Είναι ένα απόθεμα όπου τα αλλιεύματα είναι πιο χαμηλά από τα τρέχοντα αλλιεύματα, αλλά θα πρέπει να μειωθεί το ΤΑΚ και να μειωθούν οι ποσοστώσεις των συμβαλωμένων μερών που αλλιεύουν το απόθεμα αυτό. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θέλει να υποβάλει προτάσεις για το Rick and Top για να απαγορευτεί η αλία του στα διεθνή ύδατα και να καθοριστεί μια μικρή ποσόστοση σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής για την αλληλεία που θα ανακατευθύνεται σε περιοχές ε, υπό εθνική αρμοδιότητα. Επίσης, η Επιτροπή θέλει να υποβάλει προτάσεις και για τον Καρχαρία, Ρενάχ, και θα υπάρξει και μία σύσταση όσον αφορά τα παρεπίπτοντα αλλιεύματα. Αυτές είναι οι γενικές γραμμές της Επιτροπής ε, για τα αποθέματα και οι συστάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής για την ετήσια συνάντηση του 2009. θα ζητήσουμε να συνεχίσει η ΚΑΤ την εξέταση ε, της στήρησης των υποχρεώσεων όχι μόνο για τον τόνο όπως έγινε φέτος, αλλά ε, θα ζητήσουμε να γίνεται το ίδιο και για όλα τα άλλα αποθέματα τα οποία διαχειρίζεται η ΚΑΤ. όπου υπάρχουν ανησυχίες για το αν τηρούνται οι υποχρεώσεις, ιδίως όσον αφορά την υποβολή δεδομένων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ρωμέβα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα οπωσδήποτε πρώτα απ' όλα να προσθέσω και εγώ τη φωνή μου στο παράπονο στη διαμαρτυρία της κυρίας Προέδρου σε σχέση με το, θέμα αυτής της έκθεσης της υπηρεσίας ελέγχου. Είναι η δεύτερη φορά, το δεύτερο έτος ε, το, που το ζητούμε. Πέρσι Κάτι παρόμοιο συνέβη. Μα απέστειλαν μια έκθεση που δεν ήταν αυτή που ζητήσαμε και φέτο υπάρχει πάλι πρόβλημα. Έχει κάθε λόγο η Πρόεδρος και πρέπει να υποστηριχθεί αυτό το παράπονο που κατατίθεται. Διότι δεν είναι τεχνικό πρόβλημα. Υπάρχει η έκθεση αυτή, αλλά είναι, α το πω έτσι, προπολιτικό πρόβλημα πολιτική βούληση που δεν μα αποστέλνουν αυτή την έκθεση. Το δεύτερο, και επικεντρώνομαι τώρα κυρίω στην συνάντηση τη ΣΥΚΑΤ, της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Τονοειδών στον Ατλαντικό. Και θέλω να ε, επιμείνω σε αυτό σε σχέση με την ε, συνεδρίαση ε, της έκτης του μήνα. Πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η αρχή. Μια ολόκληρη σειρά ερωτήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε να διατυπωθούν. Πρώτα απ' όλα, το σημείο αφετηρίας σε σχέση με τον ερυθρόπτερο τόνο το αναγνωρίζουμε φέτος ε, υπάρχει ο κίνδυνος, ο ερυθρόπτερος ε, τόνος να πριτανεύει, να δεσπόζει κυρίως στις ε, συζητήσεις και στα θέματα. Είναι μια σοβαρή κατάσταση αυτή και νομίζω είναι αναπόφευκτο να γίνεται βέβαια κάτι τέτοιο, όμως παρόλα αυτά ενώ συμφωνώ ότι και τα άλλα είδη πρέπει εξίσου να, να σε σχέση με τον ερυθρόπτερο τόνο ε, χαιρετίζω το γεγονό ότι υπάρχει βούληση να ληφθούν υπόψη οι επιστημονικέ συστάσει. Θα θέλω όμω προ αυτό να κάνω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Την προηγούμενη εβδομάδα, όπω είπε η Πρόεδρο, είχαμε μια συνεδρίαση τη Επιστημονική Επιτροπή στη Μαδρίτη. Ήταν σαφή η σύσταση. Υλοποιούνται οι όροι και οι προποθέσει ώστε ο ερυθρόπτερο τόνο να ενταχθεί στο παράτημα 1 τη ΣΥΤΕΣ, των απειλούμενων δηλαδή ειδών όσον αφορά την απαγόρευση του εμπορίου αυτών των ειδών διεθνώς. Αυτό σημαίνει υπό την επιστημονική προσέγγιση δεν βρίσκεται άλλη ε, λύση παρά μηδενική ποσόστοση. Κάναμε λόγο ε, πέρσι για κάποιες χιλιάδες τόνους. Εφέτος, ακολουθώντας τις συστάσεις που απορρέουν από τις ε, επιστημονικές συστάσεις της προηγούμενης εβδομάδας, κατανοούμε ότι η μόνη λύση θα ήταν η μηδενική ποσόστοση. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η αξιολόγηση που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποια είναι η εντολή με την οποία θα καταλήξει στη Ρεσίφη. Η δεύτερη ερώτηση και αυτή συνδέεται επίσης με αυτή την πτυχή από ό,τι κατανόησα, το θέμα τη δυνατότητα, τη ικανότητα είναι πολύ σημαντικό θέμα και εντάσσεται και σε άλλου τομεί. Για παράδειγμα, όταν έχουμε το θέμα του κανονισμού και του ελέγχου σε σχέση με την πράσινη βίβλο, είναι εξίσου θεμελιώδε. Αλλά δεσμευόμενο με αυτό, συνδεόμενο με αυτό, έχουμε και δεσμεύσει, υποχρεώσει με συγκεκριμένε χώρε. Για παράδειγμα, για το Μαρόκο, αναφέρομαι εξειδικευμένα, σε σχέση με την ε, μείωση τη ικανότητα των δικτύων ε, των δικτύων επιφανείας ε, και για τα οποία τουλάχιστον εγώ δεν έχω επαρκή ε, εξειδικευμένα στοιχεία για το ποια είναι η κατάσταση των αποθεμάτων πόρων σε σχέση με αυτή την συγκεκριμένη κατάσταση πραγμάτων και ποιο είναι, ποιος είναι ο τελικός στόχος αυτών των δαπανών. Και αυτό είναι ένα θέμα που μέσα στο πλαίσιο συνεδρίασης της ΙΚΑΤ θα πρέπει να συζητηθεί. Και η τρίτη και τελευταία ερώτηση είναι δεν είχα ακόμα ευκαιρία να το διαβάσω βέβαια, αλλά υπάρχει η έκθεση ιδιαίτερα εξειδικευμένη και με λεπτομερή στοιχεία για την κατάσταση της εμπορίας του ερυθρόπτερου τόνου πρόσφατα και για το ε, θέμα της διεθνούς ανάλυσης ε, για αυτό το είδος. Είναι μια έκθεση που έχει συνταχθεί από την Tuna Ranching, Ranching Technologies πολύ σημαντικό για την κατάσταση στην οποία αναφερθήκαμε στην αρχή, την ευαίσθητη δηλαδή κατάσταση, την ευαίσθητη ισορροπία που αφορά τον ερυθρόπτερο τόνο. Θα ήθελα να ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πρόσβαση σε αυτήν την έκθεση και ποια είναι η αξιολόγησή τη για αυτή την έκθεση, για αυτό το περιεχόμενο. Και τελευταίο, όσον αφορά την έκθεση για την Επιστημονική Επιτροπή τη προηγούμενη εβδομάδα, Ακόμα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, δεν έχει ε, δημοσιευθεί ακόμα η έκθεση. Θέλω να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έχει, αν υπάρχει. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτήν. Ευχαριστώ. Πριν δώσω τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πω κάτι στον κύριο Ρωμέβα. Εγώ την έχω την έκθεση αυτή και την έκθεση. Δεν αληθεύουν αυτά τα οποία λένε κάποιοι. Και κάτι παραπάνω. Δεν θα σας διαβάσω την έκθεση που την έχω εδώ και την έχω διαβάσει, αλλά θα διαβάσω ένα σημείωμα που τυπώθηκε, δημοσιεύθηκε στη σελίδα του διαδικτύου σε σχέση με την συνεδρίαση 21-23. Λέει και σας διαβάζω την σελίδα. Οι επιστήμονες της ΙΚΑΤ συνήλθαν στη Μαδρίτη 21-23 Οκτωβρίου 2009 για να διατυπώσουν την αξιολόγηση στην επιστημονική από πλευρά ΙΚΑΤ για την κατάσταση των ερυθρόπτερων τόνων στον Ατλαντικό όσον αφορά τα βιολογικά κριτήρια για να συμπεριληφθεί το είδος και τα θαλάσσια είδη που εμπορικά εκμεταλλευόμαστε σε αυτό το παράδειγμα προαναγγείλαμε και απευθύναμε ε, ειδοποίηση ότι υπάρχουν μερικές και μεροληπτικές ε, ε, αναλύσεις και ερμηνείες αυτής της, αυτού του κανονισμού. Συνιστούμε οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν υπόψη συνολικά την συνολική αξιολόγηση την επιστημονική που έγινε από πλευρά μα. Δεν σα διαβάζω τίποτα παραπάνω εγώ από αυτό. Εγώ το διάβασα φυσικά και η ερμηνεία είναι σαφώ αντίθετη από αυτά τα οποία διαδίδονται και διαχέονται. Θα θέλω όμω, εν πάση περιπτώσει, να σημειωθεί η ίδια η αποσαφήνιση που έκανε η Επιστημονική Επιτροπή για τι ερμηνείε που δίνονται από πλευρά κάποιων μη κυβερνητικών οργανώσεων. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Την έχω την έκθεση από τα τρία κριτήρια υπάρχουν ε, δύο συγκεκριμένα και το τρίτο είναι η ερμηνεία σε σχέση με την ε, ΤΑΚ δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνω εγώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, έχετε, υπάρχει ικανότητα σε σχέση με τον Ερυθρόπτερο Τόνο να διαβάσετε, να κατανοήσετε. Θέλω να το αποσαφηνίσω αυτό, γιατί υπάρχουν κάποιε ερμηνείε που η ίδια η Επιτροπή η Επιστημονική τη ΣΥΚΑΤ λέει το αντίθετο. Υπάρχουν κάποιε ερμηνείε λοιπόν που στρεβλώνουν τα πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι οι ορθές ερμηνείες. Δίνω τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευχαρίστω να σας δώσω και την έκθεση. Μπορεί να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συγκεκριμένες ερωτήσεις του κυρίου Ρωμέβα, παρακαλώ. Ε, θα προσπαθήσω. Δεν θα επαναλάβω τα όσα λέει η έκθεση, γιατί υπάρχουν και στην ιστοσελίδα της ΣΥΚΑΤ μελετούμε τα πορίσματα και κάνουμε και την παραβολή με άλλες εκθέσεις. Δεν ε, έχει πολύ καιρό που εκπονήθηκε αυτή η έκθεση. Όπως είπε η Πρόεδρος, μπορεί να ερμηνεύσει κανείς με διαφορετικούς τρόπους τα πορίσματα. Διάφορα σενάρια μπορούμε να φανταστούμε. Και δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το ένα είναι πιο πιθανό από τα υπόλοιπα. Η Επιστημονική Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την κατάσταση λαμβάνοντας υπόψη αυτά που ξέρουμε και λαμβάνοντας υπόψη και την έκθεση. Για να λάβουμε υπόψη για αυτό το κριτήριο του ΣΥΤΕΣ, τη σύμβαση ΣΥΤΕΣ, για την προστασία των ειδών. Έχουμε τη βάση για την ανάλυση, αλλά σας λέω τα αποτελέσματα είναι πολλά και διαφορετικά. Στο ΡΕΣΥΒ στη Βραζιλία ε, είναι δυνατή συζήτηση με τους εμπειρογνώμενες, τον πρόεδρο του SRS. Ε, ε, ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής θα παρευρεθεί. Θα υπάρχει αντιπροσωπεία από την Επιτροπή. Διάφοροι εμπειρογνώμονες, ειδικοί για τον ερυθρό τόνο, θα διαβολευτούν για να βρούμε τη βέλτιστη δυνατή λύση. Ε, όλοι, είναι προ συμφέρον όλων μας ε, να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση το απόθωμα. Είναι καλό για μας ε, και για την βιομηχανία που εξαρτάται από την κατάσταση του αποθέματος. Αυτό είναι το εφαλτήριο για το Ντουμπρόβνικ και για το Μαρακές. Και είναι η κατάσταση τώρα. Έχουμε, επικρατεί μεγάλη αβεβαιότητα για το απόθεμα. Με κάποιο τρόπο πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Ε, τα αλλιεύματα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την κοινότητα. Πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μα είμαστε πάντω σε καλύτερη θέση σε σχέση με τον Ντουμπρόβνη και το Μαρακέ. Έχουμε περισσότερα στοιχεία σε σχέση με πέρσι. Αναφέρεται αυτό στην έκθεση. Θα γίνει ιδέουσα ανάλυση και στο μέλλον εξάλλου θα έχουμε, πώς να το πω, πιο αξιόπιστες αναλύσεις, πιο σίγουρες καλύτερα να πω αναλύσεις, διότι τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι πιο αξιόπιστα τώρα. Ε, για τα δίχτυα το, στα παρασυρώμενα πλάδια τώρα, Υπάρχουν δύο σχετικές συνεδριάσεις. Το Μαρόκο θα υποβάλει την αναφορά για, την, για τον αφοπλισμό του στόλου με παρασυρώμενα πλάδια που θα αρχίσει να ισχύει ε, από του χρόνου, αν δεν κάνω λάθος. Ε, αυτό θα συζητηθεί στο Ρεσίφι στη Βραζιλία και νομίζω ότι απάντησα έτσι σε όλες τις ερωτήσεις. Eh, Εντάξει, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και λοιπόν, ο κύριος ε, Ρωμέβα, εμένα επιμένω σε σχέση με την έκθεση αυτών που συνέβησαν στην Επιτροπή. Φυσικά υπάρχουν κάποιες ε, διαφορές σε σχέση με τις κοινοβουλευτικές ομάδες και εμάς, όμως το ε, θεμελιώδες και ουσιώδες είναι να είναι αντικειμενικά αυτά τα στοιχεία και για τον ένα και τον άλλον. Τουλάχιστον για την ερμηνεία. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνω. Και σε σχέση με την Επιτροπή διάβασα μια πληροφορία που σε σχέση με τη Μεσόγειο ε, με ενημέρωσαν ότι υπήρξαν παράπονα για τις ε, σπάνιες πληροφορίες που, οι λίγες πληροφορίες που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ερυθρόπτερο τόνο. Και αν κάποιος ενδιαφέρεται ακριβώς για τον ερυθρόπτερο τόνο, είναι οι μεσογειακοί αλληλείς που εκπροσωπούνται στην ΡΑΤ. Και εκείνοι έχουν έλλειψη πληροφόρησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θέλω να καταχωρηθεί αυτό και να αναφερθεί ακριβώς και το παράπονο ράτα της, το, της Μεσογείου. Και ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο το 5, περνάμε στο 6, σύστημα ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα αλλιέασα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού. Και πάλι είναι λοιπόν μια έκθεση που εγκρίναμε σε σχέση με την ΑΦΟ για την μεταφορά και εφαρμογή της ε, κοινοτικής νομοθεσίας συστάσεων που ελήφθη από την Ολομέλεια μιας ε, ειδική επιτροπής για την αλληλεία που έχει αυτό το ακρόνιμο. Την τελευταία φορά πάλι τα ίδια προβλήματα υπήρχαν καθυστερήσεων όσον αφορά τη μεταφορά της ε, ε, νομοθεσίας. Αυτά τα οποία ισχύουν και για την ΑΦΑ τα ίδια ισχύουν και βλέπουμε όπως και εδώ. Το συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο δεν είχαμε βρει όσον αφορά τον, την πρόταση κανονισμού της ΝΑΦΟ που εγκρίναμε προηγούμενα, είναι λοιπόν το ξεχωριστό πρόβλημα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο άρθρο 48 μέσω της διαδικασίας της επιτροπολογίας Comitology θέλει μελλοντικά όλες αυτές οι τροποποιήσεις κανονισμού Δηλαδή όλες αυτές οι προσαρμογές και εφαρμογές κοινοτικής νομοθεσίας να γίνονται μέσω επιτροπολογίας και όχι με διαβούλευση και γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Όπως ξέρετε είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται συζήτηση όχι μόνο στην Ευρωβουλή που έπρεπε να ξεκινήσουμε με πολλά νέα μέλη μετά τις ευρωεκλογέ, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο εκρεμεί και είναι σημαντικό και στο Συμβούλιο, διότι όλες αυτές οι τροποποιήσεις εξουσιών και αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων δεν είναι σαφείς υποθέσεις, δεν είναι απόλυτα σαφή πράγματα. Και με την έναρξη σε ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας αλλάζουν και τα πλαίσια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα δικαιολογεί το ότι οδηγεί αυτό στην ε, επιτροπολογία με το στόχο λέει, να, είμαστε, να είναι ταχύτερη η διαδικασία εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας και αποφάσεων που πρέπει υποχρεωτικά να ε, εφαρμόζονται και που λαμβάνονται από τις Συμβουλευτικές Επιτροπές αλλίας Αλλά η Ευρωβουλή μέχρι σήμερα πάντα έλεγε ότι αυτή η εφαρμογή πρέπει πρώτα να περνάει από την Ευρωβουλή και μετά από το Συμβούλιο όταν και σε σχέση με την συναπόφαση έτσι πρέπει να γίνεται. Αλλά και πάλι λοιπόν Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Δεν είναι πολύ πρόθυμοι όμως να δώσουν ε, αυτές τις ε, εξουσίες. Και εφόσον δεν έχουμε κάτι διαφορετικό και εφόσον δεν υπάρχει κοινό όραμα μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, θα έλεγα να μην αλλάξουν οι διαδικασίες αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό λοιπόν έχω προτείνει μια τροπολογία να διαγραφεί το άρθρο 48. Το ίδιο πρόβλημα τίθεται, είναι αυτονόητο, και στην έκθεση του συναδέλφου για ε, το Γενικό Συμβούλιο αλίας της Μεσογείου. Είναι καλό να ληφθεί μια τέτοια απόφαση, δηλαδή σε σχέση με τα τρία θεσμικά όργανα, να ισχύει αυτό μέχρι ότου ληφθεί άλλη απόφαση. Κατανοώ εν μέρη την, ε, τα επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέει ότι δεν έχει πολλά στελέχη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν έχει υλική επιμελητιακή υποστήριξη και είναι πρόβλημα να αποστέλουν το θέμα στο Κοινοβούλιο, να αναμένουν το Συμβούλιο για όλα αυτά τα θέματα. Τα κατανοώ όλα αυτά. Αλλά δεν πιστεύω ότι η αρμοδιότητα είναι να δοθούν περισσότερε ε, εξουσίε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή είναι η πρότασή μου εν αναμονή μιας μελλοντικής πιθανής συμφωνίας. Και η μόνη τροπολογία είναι για τη διαγραφή του άρθρου 48. Αυτό προτείνεται, ώστε στο μέλλον να λαμβάνονται σε σχέση με την, ε, την υπόθεση αυτή αποφάσεις ε, ε, μέσω επιτροπολογίας. Σε αυτό αναφέρεται. Αν συμφωνείτε θα δώσω τον λόγο πρώτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως θα ήθελα να σας εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους συντάξαμε αυτή την τροπολογία διαγραφής του άρθρου 48 για να είναι κατανοητό για όλους εσάς αυτό, γιατί το έκανα δηλαδή αυτό. Και έτσι δίνω το λόγο τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πιστεύω ο κ. Νούμαν είναι παρόν και την εκπροσωπή, από την Γενική Διεύθυνση Μάρα. Έχετε τον λόγο κύριε Νιού. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Νομίζω ότι σωστά εξηγήσατε τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην εισαγωγή που κάνατε. Ο σκοπός μας με το άρθρο 48 είναι να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να τροποποιούμε αυτό τον κανονισμό εγκαίρως. Όσον αφορά την ΕΑΦΚ, γίνεται η ετήσια συνάντηση τον Νοέμβριο και εγκρίνονται πολλές συστάσεις προς εφαρμογή και συνήθως αρχίζουν να ισχύουν από την αρχή της επόμενης χρονιάς. Άρα είναι πολύ πιεστικό το χρονοδιάγραμμα. Αυτές οι τροπολογίες συναντώνται στο πλαίσιο της ΝΕΑΦΚ, παρουσία των κρατών μελών, άρα δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μονομερός από την Επιτροπή. Είναι κάτι το οποίο συζητείται πλήρως με τα κράτη-μέλη. Επομένως, αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι να μπορεί η ευρωπαϊκή κοινότητα να πληρεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις και να εφαρμόζει το συντομότερο δυνατόν τα διάφορα μέτρα τα οποία εγκρίνονται σε διεθνές επίπεδο στην ΕΑΦΚ, Επιτροπή Ελίας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτείναμε την επιτροπολογία για την τροποποίηση του κανονισμού όπως κάθε φορά θα είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ. Ε, Εγώ απλά θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που είπατε ότι αληθεύει στις συνεδριάσεις ε, των ε, εκπροσωπήσεων αυτών τα κράτη-μέλη, τουλάχιστον εκείνα που, που θέλουν να παρακολουθήσουν, μπορούν να είναι παρόντα. Όμω, όχι όπω γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό το αίτημα τη Ευρωβουλή εξακολουθεί να ισχύει γιατί εμείς ως παρατηρητές συμμετέχουμε και σε μια κατάσταση ως παρατηρητές πάρα πολύ ευαίσθητη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, <clears throat> για το Συμβούλιο, από ό,τι ε, είναι ε, γνωστό, μια τέτοια, ένα τέτοιο επιχείρημα δεν εξυπηρετεί ούτε και για την Ευρωβουλή. Λοιπόν, ευχαριστώ τα σχόλια, ε, για τα σχόλια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητώ τώρα να σας παρουσιάσω το χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών καθορίζεται για τις 5 στις 17.00, ε, 5 το απόγευμα. Ψηφοφορία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 1η Δεκεμβρίου. Θα πάει στην Ολομέλεια, <clears throat> στην Ολομέλεια περίοδο συνόδου του Δεκεμβρίου. Και αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, ολοκληρώνεται και αυτό το σημείο, το 6 στην ημερησία διάταξη και περνάμε στο 7 το οποίο είναι το μακροπρόθεσμο σχέδιο για το απόθεμα <clears throat> γάβρου στον βυσκαϊκό κόλπο και για τις αλλιευτικές δραστηριότητες γάβρου. <clears throat> Η συγγήτρια είναι η κυρία ε, Μιλμπάου έχει ε, υποβληθεί σε σχέση με την τελευταία συνεδρίαση. Είχαμε εκπρόσωπο του τομέα που είχε από την εισηγήτρια προσκληθεί και χωρίς να καθυστερώ τώρα, παρακαλώ, εδώ είναι συνάδελφος, η κυρία Μπιλμπάο, θα λάβει τον λόγο η κυρία Μπιλμπάο και μετά θα λάβουν τον λόγο οι ευρωβουλευτές που επιθυμούν για να παρέμβουν σε σχέση με την έκθεση αυτή που με ιδιαίτερη ταχύτητα εμπόρεσε να συντάξει η συγγήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει η κυρία Μπιλμπάου. Πρώτα, πρώτα απ' όλα θέλω να προσθέσω και εγώ τη φωνή μου και είναι αυτονόητο αυτό στο παράπονο το οποίο εκφράσατε στην αρχή αυτής της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής Αλίας. Θέλω να υπενθυμίσω ότι, ότι αυτή η πρόταση κανονισμού Τέλη Ιουλίου είχε ε, υποβληθεί στην ε, Ευρωβουλή. Αρχίσαμε να εξετάζουμε το Σεπτέμβριο διαδικαστικά. Το χρονοδιάγραμμα που είχε προβλεφθεί, χωρίς να χάσουμε ούτε ένα λεπτό, ήταν αυτό το οποίο ακολουθούμε και τώρα. Η παρουσίαση δηλαδή και ανταλλαγή ε, απόψεων το Σεπτέμβριο, η παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης στη συνέχεια σήμερα, 3 Νοεμβρίου, Έναξη προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών, άνοιγμα προθεσμίας, 30 Νοεμβρίου, 1 Δεκεμβρίου ψηφοφορία του σχεδίου έκθεση για να ολοκληρωθεί στην Ολομέλεια του Στρασβούργου στη συνέχεια με την έγκριση. Θέλω να υπενθυμίσω εδώ κάτι. Ότι ενώ εξετάζαμε και είχαμε περάσει διαδικαστικά στην εξέταση τη έκθεση με τι προτάσει του τομέα, μάθαμε ότι θα ενέκρινε ένα κανονισμό, κανονισμό ελέγχου το Συμβούλιο, που <clears throat> θα είχε άμεσα επιπτώσει σε 14 άρθρα αυτής της πρότασης κανονισμού. Μετά από δύο λοιπόν συνεδριάσεις και αρκετές ε, εβδομάδες τηλεφωνικών επαφών καταφέραμε τουλάχιστον να μας αποστείλουν αυτήν την έκθεση για να δούμε ποια, ε, πώς θα επηρεαζόταν αυτή η ε, έκθεση σε σχέση με τον κανονισμό που ενέκρινε την προηγούμενη εβδομάδα το Συμβούλιο. Σε αυτό προστίθεται και μια άλλη νέα είδηση πάλι. Και εδώ θα ήθελα τουλάχιστον να μπορέσετε να αποσαφηνίσετε αυτό το θέμα. Γιατί εγώ σήμερα το πρωί δεν ήταν σε θέση να το διευκρινίσω, γιατί δεν είχα πληροφορίες. Πήρα μια έκθεση από την ΡΕΠΕΡ, όπου μου λένε, αναφέρεται ότι αυτή η πρόταση κανονισμού θα συζητηθεί στην ομάδα εσωτερικής πολιτικής ε, της ομάδας του Συμβουλίου και της Προεδρίας για την πολιτική συζήτηση και πιθανή έγκριση στο Συμβούλιο Αλληλείας στις 19 δηλαδή και 20 Νοεμβρίου του 2009, τρέχοντος έτους δηλαδή. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει, αν όλα αυτά αληθεύουν βέβαια, ότι το Συμβούλιο θα εγκρίνει. Αυτή είναι τουλάχιστον η πληροφορία που μου απέστειλαν. Αν κάποιος λοιπόν μπορεί να το... Συγγνώμη που σας διακόπτω κυρία εισηγήτρια, λέει η πρόεδρος. Στην ρεπέρ Ισπανική ή της Τσεχίας μπορεί κανείς να πει ότι θέλει. Το Συμβούλιο όμως δεν μπορεί να εγκρίνει τυπικά και επίσημα. Δεν μπορεί να εγκρίνει αυτή την πρόταση χωρίς να υπάρχει γνωμοδότηση του Ευρωκοινοβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν η, <laughs> η ρεπέ της Ισπανίας μπορεί να πει οτιδήποτε. Αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί έτσι χωρίς γνωμοδότηση της Ευρωβουλής. Λοιπόν, μην ανησυχείτε, δεν μπορούν να εγκρίνουν ε, κάτι χωρίς τη δική μας γνωμοδότηση. Μέχρι να έχουμε εμείς γνωμοδοτήσει δεν μπορούν να εγκρίνουν. Λοιπόν, αυτό που μου είπατε με καθησυχάζει και ελπίζω ότι θα αναμείνουν την γνωμοδότηση και την ψήφιση αυτού του κανονισμού το Δεκέμβριο από την Ευρωβουλή πριν από την έγκριση αυτής της πρότασης από πλευρά τους. Λοιπόν, τούτου λεχθέντος πρέπει να πω και κάτι άλλο. Να πω ότι καταθέσαμε τροπολογίες σε αυτόν τον κανονισμό. Δύο τροπολογίες συγκεκριμένα, θεμελιώδους σημασία για τον τομέα. Η πρώτη αναφέρεται στη σκέψη αυτού που θεωρείται ως τάκ. Δηλαδή εντάσσεται η πρόταση στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το γάβρο είναι μια πτυχή που ποτέ δεν είχε ληφθεί συνολικά σφαιρικά υπόψη. Και επιπλέον τα επιστημονικά επιχειρήματα που έχουν ε, ε, κατατεθεί και ως μνημόνιο και ως πληροφορία θα πρέπει να οδηγήσουν στο να αποκλείεται ο γάβρος από αυτές τις δυνατότητες. Τώρα, σε σχέση με τον δίκτυ ε, εκμετάλλευσης 0,3 μετά από πρόταση του τομέα και αν δεν υπάρχουν και χωρίς να υπάρχουν επιχειρήματα ενάντια από επιστημονικούς τομείς, πρέπει να είναι από το 0,3 0,4 αυτός ο δείκτης για θεμελιώδους, θεμελιώδεις λόγους. Δεν θα επαναλάβω όλες τις τροπολογίες που βρίσκονται στην έκθεση, αλλά δεσμεύομαι να αποστείλω σε όλα τα μέλη αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που έχουν επομιστεί την ανάλυση αυτού του θέματος, μία έκθεση που θα εξηγεί πώς θα επηρεαστούν τα άρθρα 8 έως 22 με την έγκριση ενός νέου κανονισμού για να μπορεί αυτό να είναι στοιχείο εργασίας για την εκπόνηση και κατάθεση τροπολογιών από πλευρά σας. Τούτου λεχθέντος θα ήθελα να διατυπώσω δύο αποσαφηνήσεις σε σχέση με την πρόταση που θέτει το Συμβούλιο, υποβάλλει το Συμβούλιο. Πρώτον, θα ήταν αναγκαίο να αποσαφηνιστεί η διαδικασία που θεσπίζεται στο άρθρο 20 της πρότασης του Συμβουλίου, το άρθρο 20, συγγνώμη, του κανονισμού του 2371, ε, ε, διότι ε, επί, συνεπάγεται ένα νέο χρονοδιάγραμμα σε σχέση με την πρόταση αυτή. Έτσι λοιπόν, για, μία, για την περίοδο αλίας μεταξύ 1ης ε, Ιουλίου και της 30ης Ιουνίου του επομένου έτους, θα πρέπει να δούμε αν αυτή η πρόταση θα, λαμβάνεται ή, θα εντάσσεται ή όχι στην πρόταση κανονισμού. Δεύτερον, θα ήταν αναγκαίο, πρέπει να πούμε, να διατυπωθεί με καλύτερο τρόπο, να διατυπωθεί, δεν ξέρω αν έχει προβλεφθεί αυτό ή όχι, σε περίπτωση που η Επιστημονική Επιτροπή δεν είναι σε θέση να υποβάλει σύσταση για τον πιο επικαιροποιημένη για το τι πρέπει να γίνει όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 αν υπάρχει πρόβλεψη για κάποια διαδικασία που θα υιοθετηθεί για να γίνεται αυτός ο υπολογισμός. Είναι ένα άρθρο το οποίο έχουμε τροποποιήσει. Είναι ένα θέμα όμως θεμελιώδους σημασία για την ανάλυση και κατάθεση τροπολογιών που έχουμε υπόψη να υποβάλουμε. Αυτά θέλω να πω και δεν θέλω να επαναλάβω κάτι, δεν θα εμείνω περισσότερο στην έκθεση. Αυτό όμως το οποίο θέλω να θέσω εν ώψη των μελών είναι, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των επιστημονικών εκθέσεων της, του φθινοπόρου, ε, θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη την πολύ σοβαρή κατάσταση που ε, διατρέχει ο τομέας ε, σε σχέση με την, ε, το πάγωμα αλληλευτικών δραστηριοτήτων και με το Ίδρυμα Άστη όσον αφορά το φθινόπωρο μας κάνει να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε σε σχέση με την βελτίωση των αποθεμάτων σε σχέση με προηγούμενα έτη. Και γι' αυτό θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσημα και τυπικά να εγκρίνουν ένα νέο τάκ ελάχιστο του επίπεδου 7.000 τόνων για το έτος 2010. Αυτό είχα να πω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριος Ρωμέβα. Σας ευχαριστώ πολύ. Απλά κάποια σχόλια και κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω εσάς, διότι πολύ γοργά, ταχύτατα, να Εντάξει, τώρα γίνεται από το αριστερό μικρόφωνο. Περιπλέκεται κάπως εδώ η διαδικασία. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για τον ταχύ τρόπο γοργά που μας υποβάλατε την έκθεση και που επικαλύπτεται, συμπίπτει και όσον αφορά τα θέματα ελέγχου ε, και οι προτάσεις που κάνει η συγγήτρια προσαρμόζονται αρκετά σε αυτά τα οποία ε, εγκρίνονται από το Συμβούλιο. Αληθεύει ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι εκείνο το οποίο εμείς επιθυμούσαμε σε σχέση με την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε σχέση με το περιθώριο ανοχής για παράδειγμα, όταν θέτει ένα 5% η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το περιθώριο ανοχής ε, συζητήσαμε στην Ευρωβουλή, καταλήξαμε στην πρόταση ότι εμείς θα θέλαμε 8% τέτοιο περιθώριο ε, το 5% εντάξει, Μπορεί να είναι και αυτό ε, λογικό. Εμείς είχαμε εγκρίνει 8, το Συμβούλιο είχε εγκρίνει 10% που είναι αυτό το οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό η πρόταση που κάνει η συγγήτρια προσαρμόζεται σε αυτά που, έχουμε ήδη, που έχουν ήδη εγκριθεί. Είναι ένα γεγονός αυτό, θα έλεγα θετικό, παρότι βέβαια θα ήταν πολύ πιο λογικό σε σχέση με την αποτελεσματικότητα και τον έλεγχο να είναι, πολύ, να είναι μικρότερο ακόμα αυτό το περιθώριο ανοχής. Το δεύτερο θέμα αφορά επίσης και το θέμα, του χρόνου πληροφόρησης ε, ε, από 4 σε μία ώρα. Προσαρμόζεται και το θέμα ελέγχου όσον αφορά το χρονικό περιθώριο. Δεν υπάρχει καμία επιπλέον ε, ένσταση, αντίρρηση. Όμως κάποιες ερωτήσεις θα ήθελα να διατυπώσω. Σίγουρα ε, δεν είχα την ευκαιρία να διαβάσω ε, κατά και εξειδικευμένα όλα αυτά. Πρώτον, ερώτηση για τον προσδιορισμό του ΤΑΚ, πράγμα το οποίο ανέφερε η συγκήτρια σε σχέση με την τροπολογία 2 για τη διαγραφή του να χρησιμοποιούνται ζωντανά δολώματα σε σχέση λοιπόν με τα, με τα τάκ του γάβρου. Μπορείτε να μας εξηγήσετε ακριβώς ε, σε τι οφείλεται αυτό και ποια είναι τα κριτήρια. Και λόγω άγνοιας ε, ερωτώ για να με πληροφορήσετε το δεύτερο στοιχείο πάλι ως ερώτηση. Συσχετίζεται και αυτό με το θέμα της διαγραφής που ε, προτείνει η, η Θα ήθελα να γνωρίζω τους λόγους, εν πάση περιπτώσει εξειδικευμένα, σε σχέση με την τροπολογία 9, που είναι μια τροπολογία διαγραφής διαγραφή σε σχέση με το γεγονός ότι στην εκφόρτωση σε σχέση με ένα τόνο ε, ε, αλλιευμάτων μπορεί να ε, υπάρχει το θέμα της έγκρισης ή μη έγκρισης. Θέλω να μπορέσει αυτό να ληφθεί υπόψη σε σχέση με αυτό το ποσό εκφόρτωσης που νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό. Δεν έχω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εσείς Η ε, κυρία Λαβίν, ευχαριστώ. Συμφωνώ με τις ερωτήσεις του κυρίου Ρομέβα και την πρόταση υπαριθμών 2. Πολύ καλό θα ήταν να μπορούσατε να μας εξηγήσετε γιατί πρέπει να αποκλειστούν τα ζωντανά δολώματα από τα ΤΑΚ. Μετά Έχω κι εγώ μία ερώτηση για την τροπολογία 5. Α. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τι έλεγε. Ότι η Επιστημονική Επιτροπή, η STCF, συμβουλεύει ότι πρέπει να κατέβουν στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο των αλλιεύμα, ε, τα αλλιεύματα και αυτό σημαίνει μείωση της τάξης του 25%. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι λίγο παράξενο, διότι μιλάμε για ένα απόθεμα που από το 2005 και μετά τελεί υποκαθεστώς κατάρρευσης, κολάψη. Και το χαμηλότερο λοιπόν επίπεδο αυτής της Επιτροπής πρέπει να είναι μηδενικό. Οπότε, εφόσον ζητείτε το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, γιατί προτείνετε μείωση μόνο 10% σε σχέση με το περασμένο έτος ε, μπορεί να μας δοθεί μια εξήγηση σε τι βασίζεται αυτή η πρόταση. Ευχαριστώ. Sí, Παρακαλώ, η Τούγκαϊθ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την εισηγήτρια, γιατί δεν μπόρεσα να είμαι παρόν στην παρουσίαση. Στην Επιτροπή Αναφορών υπήρχε ταυτόχρονη, ας το πω υποχρέωσή μου και δεν μπόρεσα να παραστώ είναι καλή φίλη μου και γνωρίζω πολύ καλά την καλή δουλειά που κάνει και ιδιαίτερα για αυτή την έκθεση για τη διαχείριση του γάβρου που είναι πολύ σημαντικό θέμα για, και για τον τομέα και για τη ζώνη γεωγραφικά από την οποία προερχόμαστε και εκείνη και εγώ στον Βυσκαϊκό κόλπο. Και είμαι βέβαιος ότι στο σύνολο η έκθεση αυτή θα είναι εξαιρετική στο σύνολο Το μόνο που θα ήθελα είναι να κάνω κάποια σχόλια Έχοντας διαβάσει προσεκτικά και την τροπολογία 5 της εισηγήτριας για το άρθρο 5, θα ήθελα να, να κατασταθεί σαφές ότι δεν θα πρέπει να είναι κατώτερο από 7.000 τόνους ε, το ελάχιστο τάκα, που είναι με σύμφωνη γνώμη του τομέα. Όμως μία ερώτηση θα ήθελα κυρίως να διατυπώσω στην Ιθάσκουν, στην Ιθάσκουν Μπιλμπάου, ιδιαίτερα δηλαδή για την έκθεση της κυρίας ε, Μπιλμπάου. Δεν θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να διευρυνθεί το μακροπρόθεσμα, μακροπρόθεσμο πρόγραμμα διαχείρισης της ζώνης 7 για να βελτιωθούν τα πράγματα. Ε, όπως όλοι γνωρίζετε ο Γαύρος ε, δεν διαχωρίζεται γεωγραφικά ακριβώς από τη μία ζώνη στην άλλη. Θα ήθελα λοιπόν σφαιρικά να λαμβάνετε υπόψη η ζώνη γεωγραφικά ως σύνολο εκεί όπου υπάρχει, υπάρχει αυτό το είδος. Με την υπερθέρμανση του πλανήτη αρχίζει να μετατίθεται περισσότερο βόρεια το είδο αυτό. Θα πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη ε, για την ε, διεύρυνση του τομέα και για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση του, της ζώνης 7. Ε, Ευχαριστώ. Πρόεδρος, λοιπόν και εγώ θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για την έκθεση της uh, κυρίας Μπιλμπάου. Λοιπόν, κυρίως θα ήθελα επίση να διατυπώσω μια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να ξεκινήσω ίσω με την ερώτηση αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπω πολύ καλά είπε η κυρία Μπιλμπάου, οργανισμός ε, ε, ανάλυσης και εξέτασης ε, σε σχέση με την διαχείριση για φέτος δημοσίευσε τον Οκτώβριο τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Είναι ενδιαφέροντα και την έχω την έκθεση. Λοιπόν, τι διαπιστώνεται. Διαπιστώνεται ότι ο γόνος που σε σχέση με το 2003 υπολογίζεται 177.000 τόνοι βιομάζα που δίνει σε σχέση με την ε, επιβίωση του αποθέματος ε, κατά την χειμερινή περίοδο υπολογίζουν μία βιομάζα ανώτερη από τις 103.000 ε, τόνους. Όπως γνωρίζετε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η πρόταση αυτή είναι η βιομάζα η προστατευόμενη σημείο αναφοράς ας το πω έτσι ως ορόσημο προστατευόμενη βιομάζα. Το στόκ, το απόθεμα εφέτος, μετά την ε, ε, διαχείριση βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Όχι μόνο όμω αυτό, η έκθεση άκτη λέει ότι είναι η ευρύτερη, ας το πω έτσι, ε, περίοδος συμμόρφωσης και σε σχέση με το 2005 και ο γόνος βρίσκεται μεταξύ των μεγαλύτερων του είδους, δηλαδή περίπου 9,5 εκατοστά, που είναι αρκετά μεγάλο. Και το απόθεμα και κυρίως τα άτομα που έρχονται σε επαφή και είναι σε επαφή με πελαγικά είδη, είναι κυκλοειδής η εξέλιξη των πελαγικών, ε, πελαγικών ειδών, έχει ανακάμψει λοιπόν το απόθεμα. Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν τώρα το απόθεμα αυτό φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και ανακάμπτει και ιδιαίτερα με την ε, ε, ανάλυση που έγινε όπως διαπιστώνετε ότι υπάρχει αυτό το στοιχείο το θετικό, καταρχήν δεν θα υπήρχε πρόβλημα για την άνοιξη, για την αλία της άνοιξης 2010, διότι είναι η καλύτερη περίοδος για την αλλιευτική δραστηριότητα αυτή. Δεν θα υπήρχε πρόβλημα λοιπόν να καθοριστεί 7.000 ε, τόνους ε, το τάκα. Όμως είναι σαφές το πρόβλημα είναι το εξής, το ακόλουθο. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να καθοριστεί τάκα από τον Ιούνιο του 2010 για την επόμενη περίοδο αλίας. Θα χάναμε δηλαδή την προηγούμενη περίοδο αλίας θα έπρεπε να είχαμε λοιπόν ένα ε, τάκ ανοιχτό, ένα, δηλαδή μια ποσόστοση ε, μέγιστου αλλιευόμενου, ε, επιτρεπόμενου συνολικού αλλιεύματος ανώτερο από αυτό, διότι έχει ανακάμψει το είδος αυτό. Δεν έχει κανένα νόημα να διασώσουμε κάτι το οποίο έχει ανακάμψει. Λοιπόν, θα ήθελα να είναι αυτό σαφές. Είναι ένα περίπλοκο θέμα. Η ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δεν θα υπήρχε δυνατότητα το Δεκέμβριο να ανοίξει ένα τάκ 7.000 τόνων με βάση την, ε, τις μελέτες ε, για την επόμενη άνοιξη αναμένοντας να εγκριθεί και να αρχίσει να ισχύει ε, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη συνέχεια. Μία, ένα σχόλιο στην, στην παρουσίαση της κυρίας εισηγήτριας. Στην τροπολογία 5, εδώ έχουμε ένα θέμα σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι στο σημείο 3. Εσείς λέτε, στην περίπτωση που η Επιστημονική Επιτροπή δεν είναι σε θέση να δώσει μια αξιολόγηση της βιομάζας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει λόγο για σύσταση για τη βιομάζα. Και νομίζω ότι έχει δίκιο σε σχέση με αυτό η Επιστημονική Επιτροπή δεν αξιολογεί τη βιομάζα. Υποβάλλει συστάσεις με βάση στοιχεία και τεκμήρια άλλων ε, οργανώσεων. Δεν αξιολογούν λοιπόν. Νομίζω η διατύπωση και η ορολογία που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η πιο σωστή. Και αυτό εδώ δεν είναι το ορθός διατύπωση. Εσείς τροποποιείτε δηλαδή σε σχέση με τη σύσταση κάτι Γι' αυτό δεν είναι ορθό. Η Επιστημονική Τεχνική Επιτροπή υποβάλλει συστάσεις, δεν αξιολογεί. Ευχαριστώ. Συνέχεια ο κύριος Κρήτον Αρσένης, παρακαλώ. Do I also have to use the other microphone? or is it because it's quite far away? No, it's okay, it's okay. Okay, they told me it's okay. So I'm going to speak in Greek. Πραγματικά συζητάμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, ένα πολύ λεπτό, πολύ τεχνικό ζήτημα ε, για το μέλλον της αλίας μια, και των αλλιευμάτων σε μια ε, σημαντική περιοχή της Ισπανίας. Ε, πραγματικά νιώθω μια σημαντική ευθύνη που έχουμε εδώ πέρα ως Επιτροπή. Ε, το μέλλον της αλίας και πολλοί από εδώ μέσα είμαστε από χώρε που η αλία είναι σημαντικό κομμάτι και τη οικονομία και των τοπικών οικονομιών. Το μέλλον τη αλία λοιπόν εξαρτάται πραγματικά από το μέλλον των αλλιευμάτων. Και πραγματικά το να προστατεύσουμε σήμερα του αλλοί σημαίνει να προστατεύσουμε και να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την βιωσιμότητα των αλλιευμάτων στο μέλλον. Ε, περίπου 2.500 οικογένειε, κάτι ένα τέτοιο νούμερο, αυτή τη τάξη είναι νούμερο, έχουν χάσει ε, πιθανόν την, την απασχόλησή του στο κομμάτι τη Αλία λόγω των, ε, ε, της κατάρρευσης των ελιωμάτων και των μέτρων που χρειάστηκαν να πάρθουν για το Γάβρο. Και αν δεν καταφέρουμε μέσα από τις αποφάσει που παίρνουμε και εδώ πέρα και στο πέρα τη Επιτροπής να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του Γάβρου, τότε θα κινδυνεύσουν ε, να υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερε απώλειες εισοδημάτων για την περιοχή, ακόμα με περισσότερε οικογένειε να, να μην μπορέσουν να συμμετέχουν ε, στην αλληλεία και να βρουν απασχόληση. Ε, ακριβώς για να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα αυτή έχει γίνει μια εξαιρετική μελέτη από το ΣΤΕΦΚ ε, και με βάση αυτή υπάρχουν κάποιες προτάσεις από την Επιτροπή. Και η δικιά μας πρόταση είναι να, να διατηρήσουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκή Επιτροπής στα βασικά της σημεία. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει να λάβει τον λόγο. Αν όχι, θα λάβει τον λόγο κυρίως ε, για να απαντήσει στις ερωτήσεις ε, των μελών. Παρακαλώ. Ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω την ερώτησή σας, Πρόεδρε, αλλά θα παρέμβω και σε μια σειρά θεμάτων που αναφέρθηκαν από την κυρία Μπιλμπάου τουλάχιστον υπάρχουν κάποιες απόσαφηνίσεις που πιστεύω ότι πρέπει να ε, τεθούν υποσυζήτηση για την δυνατότητα να ανοίξει η αλλιευτική περίοδος. Ειλικρινά αυτό το οποίο έκανε το άκτη είναι υλοποίησε μια ακουστική α το πω έτσι ανάλυση εκτίμησης της βιομάζας που υπάρχει γόνου, νέου γόνου. Τι κάνει, τι κάνει αυτή η περίοδος που δεν αποτελεί ακόμα μέρος του πρωτοκόλλου της ε, επιστημονικής ε, διατύπωσης. Εκτιμά ότι αυτή η βιομάζα είναι σε σχέση με το ε, χειμώνα ακριβώς όταν η βιομάζα των γόνων είναι υποκίνδυνο θνητότητας ε, λόγω των κλιματικών συνθήκων. Η άκτη λοιπόν σε σχέση με τις γαλλικές αρχές κάνει αυτή την ανάλυση και όταν έχει περάσει το, ο χειμώνα. Διότι έτσι έχουμε μια πολύ καλύτερη βάση, αξιόπιστη βάση όσον αφορά το απόθεμα. Και έτσι μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι η βιομάζα που είναι διαθέσιμη για την αλίευση του είδου. Μια και στο μηχανισμό, στο πρωτόκολλο, το τεχνικό μηχανισμό και πρωτόκολλο δεν εντάσσεται η ε, δράση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί ότι μπορεί να αρχίσει η αλληλευτική δραστηριότητα σε αυτή την περίοδο, όταν ακόμα απουσιάζει ένα σημαντικό στοιχείο για τις άλλες δύο, ας το πω έτσι, και τις, ε, ε, του χειμώνα και της ε, άνοιξης για να καθοριστεί η βιομάζα. Δεν θα ήταν, αυτό για να δείτε ότι θα ήταν πολύ υποκειμενικό το να πει κανείς ότι υπάρχει γόνος και βιομάζα στην θάλασσα και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει κανείς να καθορίσει μια ε, ποσόστοση 7.000 τόνων. Θα έλεγα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι και με αυτό το οποίο έχει γίνει αρκετές φορές σε σχέση με το Γάβρο για διάφορα πολιτικά επιχειρήματα αρχίζει η αλληλευτική δραστηριότητα χωρίς να είμαστε απόλυτα βέβαιοι για το απόθεμα. Η καλύτερη ιδέα λοιπόν σε σχέση με τα αιτήσια αυτά θέματα όσον αφορά το Δεκέμβριο για να έχουμε ένα αντικειμενικό πρόγραμμα, με μια αντικειμενική προοπτική, με την ακουστική ε, μελέτη, ανάλυση και με την μελέτη των οών και την, της επόασης οών γόνου. Και ιδιαίτερα όσον αφορά το χειμώνα, περίοδο που θνίσκουν οι περισσότεροι, πολλοί από τους γόνους, για να έχουμε έναν υπολογισμό αντικειμενικό για το ποια θα ήταν η αξία της βιομάζας όσον αφορά το τάκ που θα έπρεπε να ανοίξει ή να κλείσει στον κύκλο, στην κυκλική εξέλιξη ετήσια όσον αφορά το είδος. Αυτά όσον αφορά την δυνατότητα το να άρχιζε η αλλιευτική περίοδος τον Ιανουάριο, το πρώτο εξάμεινο δηλαδή του 2010 δεν ξέρω, Πρόεδρε, αν μπορώ να συνεχίσω κάνοντας ένα σχόλιο στη συνέχεια, συνεχίζοντας, διότι ευχαριστώ φυσικά την κυρία Μπιλμπάου για τη δουλειά που έκανε συντάσσοντας την έκθεσή της. Όμως, θεωρώ σημαντικό να αποσαφηνίσω κάτι εδώ. Να αποσαφηνίσω πρώτα το γεγονός ότι ότι συμπεριλάβουμε τα ζωντανά δολώματα, ιδιαίτερα όσον αφορά την, ε, το γάβρο μικρότερο του ενδεδειγμένου του ε, μεγέθους αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη του ότι στη θάλασσα υπάρχει η ε, θνησιμότητα εκείνη σε σχέση με το είδος και λαμβάνοντας υπόψη αυτή την πληροφορία και με την ε, αν δεν διαβιβαστεί αυτό το στοιχείο στην Επιστημονική ε, Επιτροπή δεν μπορεί να υπολογιστεί ακριβώς ε, η ακριβής ποσότητα. Και γι' αυτόν τον λόγο με αρκετέ αφορμές όταν αρχίζει η αλλιευτική περίοδος το ζωντανό δόλωμα, τα ζωντανά δολώματα ήταν σημαντική υπόθεση. Αλλά σε σχέση με τη διαβίβαση είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο. Τώρα σε σχέση με την τροπολογία 3 να συμπεριληφθεί η, όσον αφορά ο μήνας του Μαΐου. Σας υπενθυμίζω εδώ κάτι και νομίζω ότι εδώ και σε σχέση με τον γαλλικό τομέα και υπάρχει το θέμα της διαβούλευσης τον Μάιο έχουμε σε σχέση με την, ε, ε, την ε, κυβέρνηση της χώρας των Βάσκων το θέμα της ε, η βιομάζα, η φυστάμενη βιομάζα, η τρέχουσα βιομάζα τον Μάιο δεν λαμβάνει υπόψη την υδάτινη ε, ε, ανάλυση, ας το πω έτσι, την ανάλυση σε σχέση με τον υπολογισμό του ΤΑΚ από πλευράς των ε, γαλλικών αρχών. Και αυτό πάλι υπάρχει εδώ στοιχείο στην τροπολογία 4. Και μετά για την τροπολογία 5, για το 10% ως ανοχή. Και εδώ αποσαφηνίζω σε σχέση με αυτό ότι αυτό το οποίο έχουμε εντάξει έχουμε προβλέψει στην, που, περίπτωση που δεν θα υπήρχαν πληροφορίες ή για οποιοδήποτε λόγο δεν θα υπήρχε δυνατότητα υπολογισμού για ένα αλλιευτικό, ε, μια αλλιευτική περίοδο, η ευθυγράμμιση της τοποθέτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με, τις, ε, με τα στόκ είναι αυτό το οποίο προτείνουμε ακριβώς με τον κανονισμό σε σχέση με το μήνα Δεκέμβριο. Δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση της βιομάζας. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η αλληλευτική προσπάθεια θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά. Θα πρέπει τουλάχιστον ένα 25% να μειωθεί το τάξη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Δηλαδή ουσιαστικά αν θέλουμε να είμαστε προφυλακτική θα πρέπει να βάλουμε ένα μηδενικό ποσοστό. Αλλά μια και ευθυγραμμιζόμαστε με τα υπόλοιπα αποθέματα, ε, έχουμε αυτή την ε, ε, πρόβλεψη εδώ για το 5%. Υπάρχει και μια ολόκληρη σειρά τροπολογιών εδώ, λαμβάνοντας υπόψη την αλλαγή στο κεφάλαιο 4 που δεν θα εφαρμοζόντουσαν αυτά τα, αυτές οι διατάξεις, αναφέρομαι ιδιαίτερα στην τροπολογία 6, στην 7 στην 10 επίσης, στην 11, 12, 13 και 14. Μια και είναι άρθρα τα οποία άμεσα μέσα στον κανονισμό για τον έλεγχο ε, εντάσσονται και αφορούν τον έλεγχο. Δεν θέλω περισσότερο να μακρηγορήσω. Όμως θα ήθελα να αποσαφηνίσω κάτι. Ότι το να περάσουμε από ένα ποσοστό εκμετάλλευσης 30% από το 0,3 στο 0,4 με συγχωρείτε δικαιολογείται με την μη ύπαρξη οποιοδήποτε κινδύνου είπατε. Αυτό δεν αληθεύει απόλυτα. Μπορεί με κάποια εκμετάλλευση κάτι το οποίο δεν ήταν σημαντικό να γίνει ξαφνικά σημαντικό. Θα πρέπει πολύ προσεκτικά να αναλυθούν τα έγγραφα της ομάδας εργασίας όπου γίνεται ανάλυση του ποια είναι η ανάλυση κινδύνου σε μία περίπτωση και σε άλλη περίπτωση, από τη μία στην άλλη περίπτωση. Σε μία περίπτωση όταν μπορούμε να πούμε ότι περνώντας από το 30% στο 40% μπορεί να υπάρχει κίνδυνος. Ιδιαίτερα μπορεί να υπάρξει υπερεκμετάλλευση και έτσι να υπάρξει μεγάλος κίνδυνος ε, για την επόμενη ε, περίοδο αλίας του αλλιευτικού αποθέματος. Ευχαριστώ. Κυρία Σιγήτρια, έχετε τον λόγο τώρα εσείς. Παρακαλώ. Θα προσπαθήσω να είμαι και εγώ σύντομη, λέει η Σιγήτρια, δίνοντας τις απαντήσεις μου. Πρώτα απ' όλα, για το θέμα του ε, ΤΑΚ, για τον ορισμό των ζωντανών δολωμάτων. Μας δώσατε επιχειρήματα και πρέπει να πω ότι όλα τα οποία θα αναλύσουμε και όλα όσα έχουν αναλυθεί λαμβάνουν πάντα υπόψη, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις ε, ε, παραμέτρους του τομέα στην φυσκαϊκή και ιδιαίτερα και τη γαλλική πλευρά. Η μέθοδος που ακολούθησα και υιοθέτησα ήταν να συμπεριληφθεί σε αυτήν την έκθεση αποκλειστικά και μόνο να συμπεριληφθούν τα θέματα επί των οποίων συμφωνούσαν όλοι. Σε σχέση με κάποιες προτάσεις κάποιων τομέων υπήρχαν προτάσεις τις οποίες δεν συμμεριζόντουσαν όλοι. Αυτές δεν έχουν συμπεριληφθεί. Εντάξει, λοιπόν, τούτων λεχθέντων Ακούσατε εσείς φυσικά τα επιχειρήματα του κυρίου Πέτιερ, του αρμόδιου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του υπεύθυνου. Εγώ λαμβάνω υπόψη όχι μόνο τις απόψεις του τομέα, αλλά και τις εκθέσεις, τουλάχιστον τις γνωμοδοτήσεις των επιστημονικών φορέων. Διότι πρώτον, τα ζωντανά δολώματα δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το τάκ. Δεύτερον, αυτό το οποίο αναφέρεται είναι ότι τα στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με την αξιολόγηση της σημασίας τους είναι παλαιά στοιχεία, προηγούμενα στοιχεία, όταν ο στόλος είχε διαστάσεις που δεν έχει πια σήμερα. Δεν υπάρχουν δηλαδή σημερινά επικαιροποιημένα στοιχεία με τη συρρήκνωση του στόλου τα τελευταία χρόνια για τις επιπτώσεις και τη σημασία αυτών των ζωντανών δολωμάτων. Δεύτερον, και επιπλέον εδώ γίνεται χρήση κάποιων ε, ιδιαίτερης θνησιμότητας ε, ε ειδών. Είναι ε, ε, είδος το οποίο ε, βρίσκεται υποκίνδυνο και εδώ ένα επιχείρημα το οποίο αναφέρει ο κ. Πετιέρ, ότι δεν έχουμε στοιχεία για το πόσα ζωντανά δολώματα εδώ φορώνται. Αυτό μπορεί να είναι αντικείμενο ανάλυση για το αν θα πρέπει να ελέγχονται ή όχι τα ζωντανά δολώματα. Μια και δεν έχουμε το ότι δεν έχουμε αυτά τα ε, πληροφοριακά στοιχεία δεν είναι επαρκές επιχείρημα για να μην συμπεριλαμβάνονται τα ζωντανά δολώματα στο ΤΑΚ. Το λέω αυτό γιατί στις ποσοστώσεις που λαμβάνονται υπόψη το να πει κανεί ότι δεν είναι σημαντικό π.χ. η θνησιμότητα, σημαντικό στοιχείο για τα ζωντανά δολώματα. Και επειδή ζωντανά απορρίπτονται επίση και στη θάλασσα. Με ρωτήσατε για την τροπολογία 9 κατά δεύτερο λόγο και γιατί δηλαδή εμείς ε, θέλαμε να υπάρξει διαγραφή του κειμένου όπου αναφερόταν ότι στο αρμόδιο κράτος και τα λοιπά οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαιτήσουν το ε, ποσό αυτό το οποίο βρίσκεται ε, επί του σκάφους να μην εκφορτώνεται προηγούμενα εδώ ο τομέας φοβάται ότι μία, η καθυστέρηση μιας αδειοδότησης εκφόρτωσης μπορεί να είναι επιζήμια για την πώληση κατά την άφηξη στο λιμάνι. Για να το λάβετε και υπόψη και να το γνωρίζετε και το λέω έχοντας γνώση του τομέα. Εγώ ξέρω πώς αλλιεύεται ο γάβρος. Φεύγουν κάθε μέρα, βγαίνουν στη θάλασσα τα σκάφη, επιστρέφουν και αυτό για την πώληση του είδους εξαρτάται από την ώρα που εκφορτώνονται για την πώληση και από την ποιότητα και η ποιότητα ε, εξίσου εξαρτάται από αυτά τα στοιχεία. Όλα αυτά κάνουν τον τομέα να φοβάται, διότι, να φοβάται διότι η καθυστέρηση θα έχει επιπτώσεις και στην ποιότητα του αλλιεύματος που θα εκφορτώνεται αν υπάρχει καθυστέρηση και για την ε, τιμή του. Εδώ λοιπόν ε, λαμβάνοντα υπόψη ότι δεν υπάρχουν όρια για αυτή την αδειοδότηση, κάθε καθυστέρηση μπορεί να είναι επιζήμια. Κατά τρίτο λόγο, η τροπολογία 5. Εδώ υπάρχουν κάποια στοιχεία. Η κυρία Πρόεδρος μου έκανε μια διόρθωση. Ίσως είναι ένα λάθος στην διατύπωση, γλωσσικής διατύπωσης σφάλμα. Αλλά θέλω να πω δύο πράγματα εδώ. Πρώτον, ανοίγει πρόκειται για ένα άρθρο γενικόλογο και ασαφές. Λέει ότι στην περίπτωση που η Επιστημονική Επιτροπή δεν θα είναι σε θέση να υποβάλει σύσταση λόγω απουσίας στοιχείων επαρκώς ε, ε, αξιόπιστων, τα τάξ ε, και οι ποσοστώσεις θα είναι οι εξής, ως ακολούθω. Πρώτον, πρέπει να δούμε σε ποιες περιπτώσεις δεν θα είναι η Επιστημονική Επιτροπή σε θέση να υποβάλει μια σύσταση. Και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, να δούμε πώς μπορούμε να πούμε σε ποιες περιπτώσεις μπορεί η απουσία αυτών των στοιχείων να ε, ρυθμίζεται. Και δεύτερον, γιατί είπαμε να υπάρξει μείωση από 25% σε 10%. Διότι σε οποιοδήποτε επίπεδο, το χαμηλότερο επίπεδο το οποίο μπορεί να συστήσει η Επιστημονική Επιτροπή είναι από 0 έως 7.000 τόνους. Εμείς με βάση τις πληροφορίες θα πρέπει να προσαρμόζονται αυτά τα στοιχεία στο ελάχιστο τάκ λαμβάνοντας υπόψη την ολέθρια κατάσταση στην οποία βρίσκεται το αλίευμα πρέπει να υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Και γι' αυτό λοιπόν το 0% όπως εδώ και 5 χρόνια ισχύει θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Είναι όμως ένα άρθρο γενικόλογο και ασαφές. Προσπαθήσαμε να το συγκεκριμενοποιήσουμε πιο εξειδικευμένα. Και αν δεν υπάρχουν λοιπόν επαρκή στοιχεία πάλι δεν θα ήταν δίκαιο για τον τομέα να είναι μηδενικό το επίπεδο αλιεύματος τουλάχιστον θα έπρεπε να τεθεί το ελάχιστο, δηλαδή ως ελάχιστο 7.000 τόνοι. Απ' την άλλη πλευρά ο κύριος Σιτουργάη, σύμφωνα με το άρθρο 2 με ρώτησε γιατί περιορίζεται στη ζώνη 8 και δεν συμπεριλαμβάνεται η ζώνη 7. Αυτό είναι ένα αίτημα λοιπόν. Ένα αίτημα το οποίο κάποια ε, ένωση ή σύλλογος ε, διατυπώνει. Αυτή την πρόταση όμως δεν την κάνουμε εμείς για την ε, ζώνη αλίας είναι η ζώνη 8 αληθεύει ότι υπάρχει όριο σε σχέση με τη ζώνη 7 όπου μπορεί να ε, σε σχέση με την ε, ε, κίνηση του αλλιεύματος. Όμως δεν έχει συμπεριληφθεί αυτή η ζώνη. Όμως οι συνεδριάσει μας και μπορώ να το πω αυτό στον κύριο Πετιέρ, εγώ σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανα αυτό τον προβληματισμό. Είπα, υπάρχει αυτή η ανησυχία, να υπάρξει ανάλυση, να δούμε τι μπορεί να γίνει, να το αναλύσουμε αυτό, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα στη συνέχεια μια στιγμή. Πιστεύω ότι... Α, ο κύριος Πετιά είπε ότι το να περάσει κανείς από τον δίκτυο εκμετάλλευσης από 0,3 στο 0,4 δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν ενέχει κίνδυνο. Εγώ πιστεύω ότι στην εξήγηση που έδωσα δεν είπα σε καμιά περίπτωση και εδώ και το έχουμε και γραπτός ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Αυτό που λέω ακριβώς είναι η μορφή εκμετάλλευσης έχει συμφωνηθεί με τον τομέα και με την, ε, ε, τον τομέα αυτό εδώ και πάνω από δύο χρόνια. Το Συμβούλιο SFSR ε, Νότου, ΣΟΥΡ, είχε πει ότι πρέπει ο δείκτης να είναι 0,4. Αυτή η πρόταση βασίζεται σε σχέση με τις εκθέσεις της Επιστημονικής Επιτροπής που συμπεριλαμβάνει τον δείκτη εκμετάλλευσης αυτών που συμπεριλαμβάνει ένα εύλογο, ένα εύλογο επίπεδο κινδύνου αυξάνοντας αυτό το δίκτυ. Δεν είναι υπερβολικός ο κίνδυνος. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι αλλάζουμε το δεκαδικό. Από 0,3 το κάνουμε 0,4. Δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνο, κίνδυνος. Λέμε ότι εντάξει και ο κίνδυνος αυξάνεται. Αλλά μέσα σε αυτό το ποσοστό από το 0,3 στο 0,4 είναι ένα εύλογο ποσοστό και όχι υπερβολικό. Και με αυτό νομίζω απάντησα. Ή αν υπάρχει κάποια ερώτηση είμαι στη διάθεσή σας και παρακαλώ να μου το θέσετε για να με ρωτήσετε για να μπορέσει να επιληθεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πέρεκ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σχετικά με την έκθεση αυτή, Καταρχήν, πιστεύω ότι οι μελέτε που γίνονται καταρχήν από το ΑΣΤΗ, το Βασικό Τεχνολογικό Κέντρο Θαλάσσιας και Διατροφική Έρευνα, και οι μελέτε που γίνονται από την IFREMER, το Γαλλικό Ινστιτούτο Έρευνα για την Εκμετάλλευση της θάλασσα, που γίνονται σε άλλη εποχή του χρόνου, ε, δεν είναι αντιφατικές, είναι συμπληρωματικές και είναι απαραίτητε. Και η ΜΕΝ και η ΔΕ, νομίζω, επ' αυτού συμφωνούμε. Αυτό είναι το πρώτο. Ε, δεύτερον, όσον αφορά το αν λαμβάνονται υπόψη τα δολώματα στι ποσοστώσει, νομίζω ότι πρέπει να δούμε ε, συνολικά ε, και εδώ συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής ε, που προτείνει να λάβουμε υπόψη μας και αυτό το τμήμα γιατί ε, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται έχει κλείσει η αλία αυτού του είδους εδώ και χρόνια και επομένω είναι ένα ειδικό πρόβλημα. Δεν ξέρουμε ακριβώς προς τα που οδεύουμε, αλλά αναμφισβήτητα είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη και τα δολώματα στα συνολικότερα λιεύματα. Και θέλω να θέσω ένα ερώτημα στην Επιτροπή. Αξιολογήσατε και άλλα στοιχεία επιζήμια, στα χαρακτηρίσω, για την εξέλιξη των ηχθιδίων του γάβρου. Ε, μιλώ για τη μόλυνση και για άλλα τέτοια στοιχεία που υπάρχουν. Για να δούμε αν υπάρχουν και άλλα προβλήματα για το είδος. υπάρχουν και άλλοι λόγοι που επισέρχονται στην αξιολόγηση. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ, κύριε Εγώ θα ήθελα μόνο απλά να προσθέσω κάτι. Να πω, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι όταν κάνει λόγο στο άρθρο 5 για 25% ότι είναι το ίδιο το οποίο αναφέρεται σε άλλα αποθέματα, δεν είναι όμως τα ίδια όλα τα αποθέματα. Υπάρχουν πελαγικά και διαφορα, διαφορετικά άλλα είδη. Δεν είναι αυτό αρκετό επιχείρημα να πείτε ότι γι' αυτό το κάνατε για 25% επειδή είναι όλα ίδια. Αυτό πιστεύω εγώ. Κατά δεύτερο λόγο, ναι, συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρξουν αναλύσεις επιστημονικές. Όμως η ανάλυση άστη είναι, δίνει αρκετή ασφάλεια και βεβαιότητα ότι σε σχέση με την θνησιμότητα, αν είναι η ίδια όπως τα τελευταία χρόνια, θα εξεπερνούσε την βιομάζα την προστατευόμενη. σε σχέση με την αρχή προφύλαξης και πρόληψης, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2005 είχαμε τάκ μηδενικού επίπεδου και μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ έχουμε ένα αλίευμα που οι Ισπανοί και οι Γάλλοι που αλλιεύουν αυτό αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη κατάσταση όταν άλλοι που βρίσκονται σε ίδια ή χειρότερη κατάσταση ούτε μηδενικό ποσοστό ούτε τίποτα άλλο. Γι' αυτό πρέπει εδώ να δούμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν υπάρξει σωστή εκμετάλλευση κατά την εαρινή περίοδο του 2010 και σε σχέση με την θνησιμότητα, δηλαδή δεν είναι ένα ε, είδος το οποίο ζει επί μεγάλο χρονικό διάστημα όπως για παράδειγμα στην Ανδαλουσία εδώ λοιπόν, σε σχέση με αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη για το μέγιστο ποσοστό αλίευσης. Έχετε τον λόγο εισηγήτρια, παρακαλώ. Εγώ απλά θα ήθελα να εκφράσω από πλευράς μου ότι στη συνεργασία με το Ίδρυμα Άστη, σε σχέση και με τις εκθέσεις και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και πολλά χρόνια με αυτές τις επαφέ πιστεύω ότι είναι υπερβολικά γνωστά όλα αυτά. Αν κάτι χαρακτηρίζει την άστη είναι η αυστηρότητα του επιστημονικού ήθους και πνεύματος στην ποιότητα των εκθέσεών τους. λαμβάνοντα υπόψη σε πολλά από τα θέματα αυτά, σε σχέση και με τα θέματα της αλλιεύσης του γάβρου, όλες τις πτυχές. Αυτό είναι δεδομένο, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη συμμετοχή στην διατύπωση κανόνων εκμετάλλευσης αυτού του προγράμματος μακροπρόθεσμης διαχείρισης και εκμετάλλευσης του γάβρου. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι η έκθεση και η πρόταση που προέρχεται από το Άστι, το ίδρυμα αυτό, αν είναι, ότι είναι επιφανειακή ή ας το πω έτσι μη σοβαρή και αξιόπιστη. Έχει αυστηρό ε, επιστημονικό επίπεδο. Δούλεψε το Ίδρυμα Άστι λοιπόν με, με αυτό το πνεύμα και εμείς τις προηγούμενες εβδομάδες εργαστήκαμε με το Ισπανικό όργανο, ε, Ίδρυμα Οκεανογραφίας και με τους εκπροσώπους και από πλευρά των Γάλλων ελήφθη αυτό υπόψη. Θέλω λοιπόν να πω εδώ ότι η αξιοπιστία το επιστημονικό πνεύμα και η καλή δουλειά που κάνει το Ίδρυμα Άστι είναι κάτι που πρέπει να προασπίσω. Πρόεδρος, εντάξει, εσείς θέλετε να πείτε κάτι, να προσθέσετε κάτι, παρακαλώ. Ε, ναι, μία διευκρίνηση. Ποτέ δεν αμφισβήτησα την ποιότητα των εργασιών της αστή. Ε, είναι αδιαφυσβήτη αυτή η ποιότητα. Έλεγα απλά ότι στην αρχή του έτους καλό θα ήταν ε, να γίνει αντιπαραβολή με αυτά που μπορεί να κάνει το Ιφραμέρ. Αλλά είναι εξαιρετική ποιότητα οι εργασίες τους. Πρόεδρος, εντάξει, είναι σαφές τώρα. Προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών. 5 Νοεμβρίου και θα ψηφίσουμε στην Κοινοβουλευτική μα Επιτροπή την επόμενη συνεδρίαση 1η Δεκεμβρίου. Έτσι λοιπόν με αυτά ολοκληρώσαμε την εξέταση του σημείου 7. Περνάμε στο σημείο 8 σημερισίας διάταξης. Πολιετές σχέδιο για το δυτικό απόθεμα Σαφριδιού και για την αλληλεία του Σαφριδιού στο απόθεμά του. Ο κύριος Γκάλακερ, εισηγητής, η, Ευρωπαϊκή, Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει την πρότασή της. Στην τελευταία συνεδρίαση είχαμε και τους εκπροσώπους ΡΑΚ πελασγικών ειδών, ο κύριος Ντόνοβαν που μας εξήγησε. Ο κύριος Γκάλακερ αποχώρησε, όχι έτσι, εντάξει, συγγνώμη. Ε, μας εξήγησε τις απόψεις ε, της ομάδας για την πελαγική αλία. Δίνω αμέσως τον λόγο στον κύριο εισηγητή Γκάλαγκερ. Uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Φαντάζομαι ότι στο Κοινοβούλιο θα έχουμε όλο και μεγαλύτερη εξουσία τώρα που και 27 χώρε υπογράφουν τη συνθήκη τη Λισαβόνα και ο πρόεδρο Κλάου νομίζω υπέγραψε. επομένω, όλα αυτά ε, είναι καλέ ειδήσει και για την Επιτροπή Αλίας γιατί αυξάνονται οι αρμοδιότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σχετικά και με την απάντηση τη Επιτροπή για το αν θα πρέπει να το καθυστερήσουμε μετά τη Λισαβόνα ή όχι, νομίζω θα έχουμε καλή συνεργασία και θα μπορούμε να το κάνουμε το Σεπτέμβριο. Η πρόταση αυτή δημιουργεί ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για το δυτικό απόθεμα ε, σαφριδιού. Ο στόχος της πρότασης αυτής είναι να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να εκμεταλλευόμεθα τους πόρους με βιώσιμο τρόπο με συνθήκες σωστές και περιβαλλοντικά και οικονομικά. Η πρόταση αυτή είναι μια πρόταση που έχουμε από τον Απρίλιο του 2009 και βασίζεται στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Αηφόρο Ανάπτυξη του 2002 στο Johannesburg. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να διατηρήσει και να αποκαταστήσει τα αποθέματα σε επίπεδα που να μπορούν να διασφαλίσουν ότι θα έχουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση και είναι μια πρωτοβουλία την οποία χαιρετίζουν οι εμπλεκόμενοι και το Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο και ο κ. Ντόναχιου τόνισαν ότι αντικατοπτρίζει η πρόταση της Επιτροπής μια ευπρόσδεκτη πρωτοβουλία. Υπάρχουν πολλοί τομείς που αναφέρονται στην πρόταση αυτή. Δεν θα, τους Δεν θα αναφέρω όλους τους τομείς. Ε, το 4α, το δελτα 2 το 4βγ, το 3α. Ε, λαμβάνεται υπόψη πάντως η Βόρειος Θάλασσα δυτικά της Ιρλανδίας, ε, το δυτικό τμήμα της ε, ε, Μάχης και το βορειοδυτικό τμήμα της Ισπανίας. Αν δούμε το χάρτη, το δυτικό απόθεμα καλύπτει το μεγαλύτερο, τη μεγαλύτερη περιοχή. Επομένως, από οικονομικής πλευράς είναι το πιο σημαντικό απόθεμα σαφριδιού. Υπάρχουν και άλλα αποθέματα, μικρότερα και εξίσου σημαντικά βέβαια. Το απόθεμα, η βιομάζα του αποθέματος αναπαραγωγής δεν μπορεί να μετρηθεί εάν έχουμε επιστημονικά δεδομένα ανεπαρκή. Κάθε τρία χρόνια όμως διεξάγονται διεθνείς έρευνες οτοκίας, όμως τα δεδομένα δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε μία πλήρη αξιολόγηση. Απουσία τέτοιων στοιχείων και χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες από τις έρευνες οτοκίας, μπορούμε, χωρίς να έχουμε τα ιδανικά στοιχεία, αλλά μπορούμε να εκτιμήσουμε τη σχετική διαθεσιμότητα του αποθέματος. Αυτή η πρόταση λοιπόν μιλά για τις δυσκολίες που υπάρχουν και διατυπώνει ένα νέο τρόπο απόφασης σχετικά με το σύνολο επιτρεπωμένων αλλιευμάτων. Και πιστεύω ότι χρησιμοποιώντας αυτό τον τύπο έχουμε υψηλή πιθανότητα μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του αποθέματος αυτού. Το 2004 κάποια ερευνητικά προγράμματα επιβεβαίωσαν προηγούμενες υποθέσεις ότι η κατανομή του αποθέματος καλύπτει τα ύδατα της βορειοδυτικής Ισπανίας και η Επιτροπή προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τους τομείς διαχείρισης που έχουν οριστεί για τον καθορισμό των ΤΑΚ. Η τωρινή θέση για τη διαχείριση δεν είναι ε, η καλύτερη δυνατή για τη διαχείριση του αποθέματος του σαφριδιού και γι' αυτό επειδή υπάρχει έλλειψη πληροφοριών, θα πρέπει να καθορίσουμε ένα τύπο για τα σκάφη που ασχολούνται με την αλία του σαφριδιού στις διάφορες περιοχές και αυτός ο τύπος βασίζεται στους καλύτερους διαθέσιμους επιστημονικούς και βιολογικούς δείκτες. Υποστηρίζω λοιπόν καταρχήν την πρόταση της Επιτροπής και θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντική η καλή συνεργασία μεταξύ του τομέα και των επιστημόνων και ακριβώς με βάση αυτή την καλή συνεργασία εκπονήθηκε και το σχέδιο. Λόγω των περιορισμένων γνώσεών μας σχετικά με τη βιομάζα του αποθέματος αναπαραγωγής, το σχέδιο χειρίζεται τα δεδομένα και τις δυσκολίες εκτίμησης με ορθολογικό τρόπο. Πιστεύω λοιπόν ότι το σχέδιο αυτό είναι καλό και προσφέρει σταθερότητα στη βιομηχανία. Έχω ήδη κάνει κάποιες προτάσεις τροπολογίας. Καταρχήν διότι οι περιοχές αποθεμάτων δεν συμπίπτουν με τις περιοχές για τις οποίες έχει οριστεί σύνολο επιτρεπωμένων αλλιευμάτων, τάκ δηλαδή. Λόγω αυτής της αναντιστοιχίας είναι απαραίτητη η προσαρμογή. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει το πρόγραμμα, καθώς εξελίσσονται οι επιστημονικές γνώσεις, θα πρέπει να δίδει τη δυνατότητα προσαρμογής των σημείων αναφοράς. Και όταν δεν μπορούμε να υπολογίσουμε επιστημονικά τα στοιχεία αυτά, επειδή είναι ευαίσθητα τα δεδομένα, και ο εκπρόσωπος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Πελαγικών ε, Ειδών συμφωνεί με αυτό το θέμα. Έχουμε υπολογίσει το επίπεδο των απορρίψεων σε 15 ετή περίοδο και θα ήθελα να προτείνω μια περαιτέρω μεθοδολογία που προτείνει τώρα και η Επιτροπή. Να λάβουμε δηλαδή υπόψη τα ιστορικά δεδομένα που έχουμε για τα τελευταία 15 χρόνια και όπως είπε ο εκπρόσωπος του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Πελαγικών Ειδών, το 5% φαίνεται ε, πολύ ψηλό και επειδή κάθε χρόνο το ποσοστό τα τελευταία 15 χρόνια ήταν κάτω από 1% και μερικές χρονιές ήταν και κάτω από 0,5%. Το μόνο έτος ε, που ήταν σχετικά υψηλό ήταν το 1996, αλλά έκτοτε ήταν σχετικά χαμηλό. Γι' αυτό έχω προτείνει μια τροπολογία σε σχέση με αυτό. Ελπίζω ότι οι επεξηγηματικές δηλώσεις είναι αρκετά απλές, ώστε να γίνουν κατανοητές από όλους και ε, προτείνω τα γενικά μέτρα ε, ελέγχου και επιτήρησης που αναφέρονται και στο πλαίσιο της απόφασης που έλαβε το Συμβούλιο Λίας στο Λουξεμβούργο την περασμένη εβδομάδα. Ε, φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα λυθούν υπόψη. με σκοπό να έχουμε σωστά δεδομένα και σωστή υποβολή εκθέσεων. Επίσης και τα σκάφη τα οποία αλλιεύουν σε μία περιοχή θα πρέπει να μπορούν ε, να ε, εκφορτώνουν ε, τα αλλιεύματά τους σε άλλη περιοχή και υπάρχει γενική υποστήριξη πέρα αυτού, δηλαδή αν αλλιεύει κάποιο σκάφο σε περιοχή όπως το 4Β να μην μπορεί να εκφορτώσει σε άλλη περιοχή που μπορεί να έχει καλύτερη τιμή για το σαφρίδι. Σύμφωνα με τους κανονισμούς θα είναι δυνατόν να γίνει αυτό αφήνοντας τα λιευτικά εργαλεία μέσα στο σκάφος και κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα έχει δυνατότητα το σκάφος να λιεύει σε περιοχή όπου δεν έχει άδεια. Έχω και κάποιες τεχνικές τροπολογίες ε, ίσονο σημασίας, αλλά είναι πολύ τεχνικού χαρακτήρα και θα υποβληθούν πριν ολοκληρωθεί η προθεσμία για τις, τροπολογίες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω το έργο που επιτέλεσε ο εισηγητής. Συμφωνώ με αρκετά από τα θέματα που παρουσιάστηκαν. Πρώτα απ' όλα <clears throat> για την ιδιομορφία που υπάρχει σε σχέση με την Ισπανία. Σε σχέση, για παράδειγμα, με το σαφρίδι, το οποίο είναι προς κατανάλωση. <clears throat> Δεν είναι ένα θέμα το οποίο ε, έχει, να έχει εξεταστεί στην προσέγγιση αυτή και σε σχέση με μια συγκεκριμένη αιτιολογική σκέψη θα πρέπει νομίζω να υπάρξει κάλυψη αυτού. Είναι σημαντικό στοιχείο. Και από πλευρά του εισηγητή καθορίστηκε πώς οι ζώνες που πρέπει να καθορίζονται και ότι σε σχέση με κάποιες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουμε ποιες είναι εκείνες οι ζώνες που πρέπει να τεκμηριώνονται ω ζώνε αλίευσης, μελλοντικέ ζώνε αλίευσης. Θα ζητούσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει και να καθορίσει αυτέ τι ζώνε, διότι μα ανησυχεί αυτό το θέμα για την πιθανή διαστηριότητα αλίευσης, αλία σε αυτέ τι ζώνε. Πρέπει να ξέρουμε ποιε ζώνε είναι αυτέ. Και υπάρχει εδώ αυτή η απουσία αυτών των στοιχείων. Θέλω να συμπληρώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μα δώσει τα συμπληρωματικά αυτά στοιχεία εδώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρο. ευχαριστώ. Άλλοι θέλουν να παρέμβουν. Ο κύριο Λεβί, παρακαλώ. Ε ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον εισηγητή. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσία. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε υποβάλει μια πρόταση για τις απορρίψεις ε, και τον τρόπο υπολογισμού τους και μιλάτε για ποσοστό όχι κάτω του 5%. Αυτό βασίζεται σε αξιολογήσεις που έχουν γίνει από επιστήμονες τα τελευταία πέντε χρόνια για τις απορρίψεις. Μπορεί να αιτιολογήσει την πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορώ να φανταστώ ότι μιλώντας για τις απορρίψεις στη θάλασσα, υπάρχει και μεγάλος παράγοντας ε, αβεβαιότητας. Είναι πολύ δύσκολο για μας να εποπτεύουμε με υφόρο τρόπο τα αποθέματα. Μπορείτε να μας πείτε πώς ακριβώς, ε, γιατί υποβάλλεται αυτή την πρόταση για την ε, καταμέτρηση των απορρίψεων. Ευχαριστώ κυρία Λεβίν. Θα ήθελα να κάνω και εγώ μια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την απολογία 10 για την έκθεση, της έκθεσης. Ερωτώ, αυτό το άρθρο 11 μπορεί να εφαρμόζεται σε σκάφη τρίτων χωρών σε σχέση με την πρόταση του εισηγητή. Έχω αμφιβολίες, αλλά θέλω να μου το επαληθεύσετε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να εφαρμόζεται και σε σκάφη τέτοια. Αλλά θέλω να μου πείτε, νομικά μπορεί να γίνει αυτό. Και μετά ένα άλλο θέμα, το οποίο θα ήθελα να, εδώ να αποσαφινιστεί. Κατανοώ ότι σε σχέση με τις τροπολογίες, την 9, την 12, την 13, που αναφέρονται στον κανονισμό, θεμελιώδη κανονισμό ελέγχου που εγκρίθηκε, όμως όλα τα προγράμματα μπορούν να έχουν δικά τους ε, μέτρα ελέγχου, αλλά πιο περιοριστικά ή όχι σε σχέση με τον κανονισμό, θεμελιώδη κανονισμό. Δεν είμαι υπέρ κατά των προτάσεων που διατυπώνονται εδώ. Στρέφομαι στο ε, να δούμε το ότι δεν συμμερίζομαι την αξιολόγηση ότι επειδή υπάρχει βασικός κανονισμός, τα συγκεκριμένα προγράμματα ανάκαμψης ή οποιαδήποτε άλλα δεν μπορούν να έχουν ειδικά μέτρα και ε, κανονισμούς ε, και διατάξεις ελέγχου. δεν θέλω να πω αν κάτι δεν είναι σωστό ή όχι, αλλά για παράδειγμα για κάποιες τροπολογίες όπως την 9 ή για την 12 και την 13 είναι ένα σχόλιο γενικού χαρακτήρα. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον κύριο Λίντερμαν της Ευρωπαϊκή Επιτροπής για να απαντήσει σε ερωτήσεις που διατυπώθηκαν και για τα σχόλια που μπορούν να γίνουν σε σχέση με την έκθεση του εισηγητή και μετά θα ολοκληρώσει ο κύριος Γκάλαχερ εισηγητής. Η Επιτροπή, ο κύριος ε, Λίντερμαν έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να πω... Ε, Καταρχήν θα ήθελα να ε, απαντήσω στα ερωτήματα που έθεσε ο κύριος Γκάλεχερ. Είναι ε, ερωτήματα τα οποία τίθενται και από τον κλάδο και από την παρουσίαση που έγινε εδώ στο κύριο του από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Πελαγικών Ειδών. Αντικατοπτρίζουν και τις ανησυχίες της βιομηχανίας. Ο δεύτερος τομέας στον οποίο ε, υπέβαλε τροπολογίες ο κύριος Γκάλεχερ, αφορά ε, το νέο σύστημα, το νέο κανονισμό ελέγχου και από αυτόν θα ήθελα να απαντήσω. Καταρχήν όσον αφορά τα ερωτήματα ε, της Επιτροπής για την προσαρμογή των στοιχείων στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Είναι απαραίτητο να το έχουμε αυτό για να μπορεί να λειτουργήσει το πρόγραμμα. Καλύπτεται ε, το απόθεμα του Δυτικού Σαφριδιού και ε, οι επιστημονικές επιτροπές ε, το προσδιορίζουν με βάση επιστημονικές μελέτες που γίνονται τα τελευταία χρόνια και είναι διαφορετικά τα στοιχεία που έχουμε τώρα σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια. Θέλουμε να βρούμε και για τα αποθέματα ε, σαφριδιού και που να βασίζεται και στα προηγούμενα δεδομένα και συγκεκριμένα αυτό σημαίνει ότι μια ε, ζώνη όπως η 8ΣΕ για την Καταβρική θάλασσα στη βόρειο, στα νυχτά της βορειοδυτικής Ισπανίας είναι μια ζώνη που μπορεί να είναι ε, μια ιδιαίτερη ζώνη ΤΑΚ χωριστή σε σχέση με την υπόλοιπη ε, δυτική ζώνη Σαφριδιού όσον αφορά ε, το πολιτές πρόγραμμα. Υπάρχει επίσης ε, και η ζώνη της Ανατολικής Μάχης που ανήκει στην περιοχή του αποθέματος της Βορείου Θαλάσσης και οι δύο αυτέ ζώνες, δηλαδή και η Ανατολική Μάχη και η Καταβρική Θάλασσα, έχουν σημαντικά αποθέματα και είναι πολύ σημαντικό να συμφωνήσουν όλα τα κράτη-μέλη με τη διαδικασία την οποία προτείνουμε. Και υπάρχει και μια μικρή προσαρμογή που πρέπει να γίνει στη βόρεια, ε, στο βόρειο τμήμα της Βορειού Θαλάσσης ε, σχετικά με το απόθεμα. Είναι μια ζώνη που ανήκει στο τάκ της Βορείου Θαλάσσης και ε, αυτό το κομμάτι της, στο βορρά της Βορειού Θαλάσσης μπορεί να συμπεριληφθεί στο δυτικό απόθεμα Σαφριδιού. Ήδη εδώ και δυόμιση χρόνια συζητούν τα κράτη-μέλη στο Συμβουλίο τα θέματα αυτά και έχουν ε, ανταλλάξει επιχειρήματα και έχουν διατυπωθεί διάφοροι τύποι για, την, ε, για τον υπολογισμό ε, των ΤΑΚ και αυτοί οι τύποι που προτείνονται νομίζω ότι τώρα πλέον ε, έχουν οριμάσει και μπορούμε πλέον να καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα φέτος. Είναι μια μακρά διαδικασία, χρειάζεται πολλή χρόνο για να οριμάσουν τα θέματα και να ληφθεί η απόφαση, αλλά νομίζω ότι τώρα μπορούμε να προωθήσουμε αυτό το πολιετές πρόγραμμα, νομίζω ότι φέτος μπορούμε να τα καταφέρουμε και στη συζήτηση έχουν προκύψει ενθαρρυντικά μηνύματα από τα κράτη-μέλη και στον ε, κανονισμό για τα τάκ και τις ποσοστώσεις για την επόμενη χρονιά θα μπορέσουμε πλέον να έχουμε αυτή τη συμφωνία, αυτά δηλαδή που θα αποφασιστούν ε, τον Δεκέμβριο. Τώρα όσον αφορά τον υπολογισμό των απορρίψεων, θέλω να πω ότι υπάρχουν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις τα τελευταία χρόνια σχετικά με τον υπολογισμό των ε, απορρίψεων και όπως είπε ο εισηγητής, είναι πολύ μικρά τα ποσοστά απορρίψεων. Όμως μερικές φορές ε, μπορεί οι επιστήμονες να μην ε, εμπιστεύονται τα δεδομένα απορρίψεων μια συγκεκριμένη χρονιάς. Και σε άλλες περιπτώσεις, ε, όταν δεν μπορούν οι επιστήμονες να δώσουν κάποια δόση, κάνουμε κάποια τροποποίηση στον τρόπο υπολογισμού και εδώ προτείνει η Επιτροπή τουλάχιστον 5% να αφαιρεθεί ο, ο κύριος Γκάλαχερ είπε ότι μόνο το 1996 ήταν σχετικά υψηλές ε, οι απορρίψεις κάτω από 5% και βάσει της αρχής της προφύλαξης ε, θα έπρεπε ε, να λάβουμε υπόψη μας αυτά τα στοιχεία που έχουμε για, τις, για την αφαίρεση από τις απορρίψεις. Από τα τελευταία 15 ε, χρόνια ε, ε, βλέπουμε ότι οι μέσες απορρίψεις είναι σχετικά χαμηλές και αν κάποια χρονιά οι επιστήμονες δεν μπορούν να δώσουν σωστά επιστημονικά δεδομένα, θεωρούμε τις απορρίψεις υψηλότερες, χωρίς όμως να το γνωρίζουν αυτό επακριβώς οι επιστήμονες και γι' αυτό εφαρμόζουμε την αρχή της προφύλαξης και δεν θέλουμε να έχουμε μόνο 0,8%. Ε, στη συνέχεια, Πρόεδρε, μιλήσατε για το ε, αν υπάρχουν διατάξεις ελέγχου για σκάφη τρίτων χωρών. Είναι δυνατό να ισχύει αυτό. Είναι δυνατόν σκάφη τρίτων χωρών στην περίπτωση του δυτικού αποθέματος αφριδιού να λιεύουν όπως στις ε, νήσεις Φερόες και στην Ορβηγία και μπορεί να έχουν πρόσβαση στο, απόθεμα, στο δυτικό απόθεμα σαφριδιού και επομένως η πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών θα πρέπει να υπόκειται σε συγκεκριμένα μέτρα ελέγχου. σύμφωνα με τη Συμφωνία για την πρόσβαση σε αλλιευτικούς πόρους. Και στην περίπτωση της προτάσεως του κυρίου Γκάλαχερ, όταν είναι υποχρεωμένα τα ε, ε, σκάφη τα οποία έχουν αλλιεύσει σαφρίδι σε άλλα ύδατα και ε, εισέρχονται στη ζώνη του δυτικού αποθέματος σαφριδιού, θα πρέπει να εφαρμόζουν τις διατάξεις τις οποίες έχουμε προτείνει και πιστεύουμε ότι είναι λογικό να εφαρμόζουν και τα σκάφη των τρίτων χωρών αυτές τις διατάξεις. Όσον αφορά τώρα τον ε, κανονισμό ε, ελέγχου, οι προτάσεις ε, του εισηγητού αφορούν τον κανονισμό και την μεταρρύθμιση του Συμβουλίου του Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τις προτάσεις, αφαιρούνται από το πρόγραμμα οι έλεγχοι που ρυθμίζονται στον Γενικό Κανονισμό Περιελέγχου δεν θα μπω σε λεπτομέρειε τώρα, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν τους ή άλλους ε, στου κανονισμού ε, περιελέγχου και έχουμε υποσχεθεί και στη βιομηχανία αλλά και στα κράτη-μέλη ότι αυτός ο κανονισμός θα συμπεριλαμβάνει πολλά ε, τμήματα και οι διατάξεις για τον έλεγχο στα πολιετή προγράμματα μπορούν να είναι συντομότερες αν έχουν ρυθμιστεί από τον κανονισμό ελέγχου και αυτά τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν στα πολιτική προγράμματα ελέγχου θα είναι οι ειδικέ διατάξεις που θα αφορούν συγκεκριμένες συνθήκες ε, υπό τις οποίες διεξάγεται η αλία. Συγκεκριμένα δηλαδή θέματα τα οποία δεν έχουν μπορέσει να επιληθούν στο Γενικό Κανονισμό ε, περί ελέγχου. Και είμαστε ανοιχτοί στην προσαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων. Εδώ, επειδή πρόκειται για πολιετές πρόγραμμα, τα κράτη-μέλη ε, είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν ε, ε, πρόγραμμα ελέγχου και είναι υποχρεωμένα τα κράτη-μέλη να υποβάλουν αυτά τα σχέδια. Θα πρέπει στο μέλλον να βελτιωθεί ο έλεγχος του δυτικού αποθέματος Σαφριδιού και αντίστοιχο πρόγραμμα υπάρχει και για τον μπακαλιάρο και αυτό θα πρέπει να γίνει και για το σαφρίδι. Θα πρέπει δηλαδή να ισχύσουν αυτά τα οποία αποτελούν γενικευμένη πρακτική. Νομίζω ότι απάντησα στα βασικά ζητήματα με αυτά που σας είπα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις εξειδικευμένες ε, σε βάθος ε, πληροφορίες. Ο εισηγητής έχει τώρα τον λόγο παρακαλώ για να ολοκληρώσει. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε σχέση με τα ύδατα βορείου της Ισπανίας, νομίζω ότι ε, έχει φροντίσει το θέμα η Επιτροπή με το νέο κανονισμό για την εποπτεία και τον έλεγχο. Είναι σημαντικό, βέβαια, να δούμε τι θα γίνει με τις τρίτες χώρες. Αν εισέλθουν συμφωνία ε, οι τρίτες χώρες για το δυτικό απόθεμα πρέπει να συμμορφωθούν με τις απαιτήσει. Ο κανονισμός για τους ελέγχους θα πρέπει να δούμε αν θα λάβει την πολιτική συγκατάθεση του Συμβουλίου του Νοεμβρίου και πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να φέρουν τις ίδιες ευθύνες και οι τρίτες χώρες αν συμμετάσχουν στη συμφωνία. Δεν αναφέρεται ρητά, αλλά Πιστεύω ότι όλοι κατανοούν ότι αυτό πρέπει να ισχύει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκάλαγε. Απλά να σας πω ότι προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών θα λήξει στις 5 Νοεμβρίου 17.00. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας την 1η Δεκεμβρίου και θα περάσει για να ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Έτσι ολοκληρώσαμε τώρα την ημερήσια διάταξη. Την εξαντλήσαμε όπως προβλεπόταν για σήμερα. Απομένει ένας συντονιστής που λείπει για να προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε τη συνάντηση των συντονιστών και λίγο πιο πριν από ό,τι προβλεπόταν, πέντε και τέταρτο. Λείπει όμως ένας συντονιστής. Έχει ενημερωθεί και θα φτάσει. Είπε θα φτάσει το δυνατόν νωρίτερα. Λέω λοιπόν να είναι παρόντες ώστε όταν θα έρθει ο απόν συντονιστής να ξεκινήσουμε αμέσως με συνεδρίαση. Εδώ διακόπτεται η λίγη συνεδρίασή μας και να παραμείνουν οι συντονιστές και όταν θα έρθει ο απόν συντονιστής θα ξεκινήσουμε με τη συνάντηση συντονιστών. Συνεδρίαση αύριο στις 9.00. ευχαριστώ.